και τώρα θέλω να δώσω το λόγο αμέσως στον πρόεδρο Μπαρόζο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, κύρια Πρωθυπουργέ Θόνινγκ Σμιτ, αξιότιμα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Θα ήθελα καταρχάς να σας ευχαριστήσω κύριε Πρωθυπουργέ για την εναρκτήρια ομιλία σας η οποία μας ε, εξέθεσε το όραμά σας για μια ενωμένη ισχυρή Ευρώπη. Όταν συναντηθήκαμε στην Ευρώπη σύντομα μετά την εκλογή σας τον Οκτώβριο πέρσι, σας είπα ότι η πεποίθησή μου είναι ότι η Δανία θα είναι αποφασιστικής σημασίας για το κοινό μας πρόγραμμα. Ακούγοντάς σας σήμερα και τις εμπνευσμένες σας παρατηρήσεις για τις ειλικρινείς ευρωπαϊκές αξίες και την κοινοτική μέθοδο, είμαι ακόμα πιο πεπισμένος για αυτό που σας είπα. Αξιότιμα μέλη, γνωρίζουμε όλοι ε, πόσο δύσκολε είναι οι οικονομικέ πραγματικότητε στην Ευρωπαϊκή Ένωση σήμερα. Τον Οκτώβριο πέρσι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε έναν ο χάρτη πέντε σημείων για την ε, ανάπτυξη και τη βιωσιμότητα. Είπαμε ότι θα πρέπει ταυτόχρονα να συνεργαστούμε για να ανταποκριθούμε στι δυσκολίε τη Ελλάδο, να ενισχύσουμε ε, την Ευρωζώνη για την αντιμετωπίση την κρίση, για να ενισχύσουμε το τραπεζικό σύστημα μέσω της επανακεφαλαιοποίησης κυρίως, να προωθήσουμε την ανάπτυξη και τη σταθερότητα και τις κατάλληλες πολιτικές και να έχουμε μια εύρωστη οικονομική διακυβέρνηση. Θα πρέπει να είμαστε σαφείς. Χωρίς την εφαρμογή ε, μιας αξιόπιστης απάντησης ε, στην κρίση της Ευρωζώνης, η οικονομική μας ευρωστία δεν θα μπορέσει να επιτευχθεί. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή λοιπόν προτρέπει τα κράτη-μέλη ε- να εφαρμόσουν αυτά τα οποία εκκρεμούν ακόμα στον οδικό χάρτη για τη λύση της Ελλάδος, για την εφαρμογή ενός αξιόπιστου συστήματος ασπίδων και όταν δημιουργήσουμε αυτό το σύστημα θα μπορέσουμε να απαντήσουμε με πειθαρχία και κυρώσεις. Χρειάζεται πειθαρχία, ναι, αλλά χρειαζόμαστε και σύγκληση. Χρειαζόμαστε σταθερότητα, είναι απαϊκανή και αναγκαία συνθήκη, αλλά χρειαζόμαστε και ανάπτυξη. Η Ευρώπη χρειάζεται περισσότερη σύγκληση, αλληλεγγύη και ανάπτυξη. Όλο και περισσότερο οι εταίροι μας και οι διεθνείς επενδυτές ζητούν ε, και ρωτούν το εξής ερώτημα. Ποια είναι το μεσοπρόθεσμο και το μακροπρόθεσμο πρόγραμμα της Ευρώπης για την ανάπτυξη. Είναι σαφές ότι δεν θα μπορέσουμε να υπερχεράσουμε την κρίση αν δεν απαντήσουμε στο ερώτημα της ανάπτυξης. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εδώ και χρόνια σας λέει τι πρέπει να γίνει. Αλλά θα πρέπει να είμαστε ειλικρινεί. Η δράση από πλευρά κρατών μελών είναι άνηση και σε κάποιες περιπτώσεις και ανεπαρκής. Εάν λοιπόν θέλουμε πραγματικά να ξεπεράσουμε την κρίση, θα πρέπει να είμαστε σοβαροί και να αναλάβουμε αποφασιστική δράση για να έχουμε ανάπτυξη ε, και να προχωρήσουμε να συμβαδίζει με την αποφασιστική δράση που έχουμε εδώ για να παραγω... Ε, ήδη εν εξελίξει για να έχουμε δημοσιονομική ένωση. Επειδή Λοιπόν, το χρειαζόμαστε. Τα κράτη-μέλη θα πρέπει να έχουν διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις για να μπορέσουμε να βοηθήσουμε τι επενδύσει και την ανάπτυξη. Πρέπει να επενδύσουμε σε προγράμματα προτεραιότητα, ιδίω προγράμματα καινοτομία. Να έχουμε τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα από κονδύλια τα οποία δεν έχουν δαπανηθεί ακόμα και να έχουμε πρόσβαση στην αγορά σε αναπτυσσόμενες οικονομίε εκτό Ευρώπη. Α δούμε και την πραγματική οικονομία και εν είδη παραδείγματος να σας πω το εξή έχουμε χονδρικά 23 εκατομμύρια ανέργους στην Ευρώπη και κατά μέσο όρο 23 εκατομμύρια μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Εάν δημιουργήσουμε λοιπόν τις κατάλληλες προϋποθέσεις για κάθε μικρομεσαία επιχείρηση ώστε κατά μέσο όρο να δημιουργήσει μία θέση εργασίας θα μπορέσουμε να πατάξουμε την ανεργία. Η απάντηση λοιπόν, η απάντηση στην ανάπτυξη βρίσκεται σε επιχειρήσεις μας, συμπεριλαμβανομένων και των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Και ο τρόπος να επιτύχουμε το στόχο αυτό είναι μέσω πιο ευέλικτων και ανταγωνιστικών αγορών, λιγότερης γραφειοκρατίας, καλύτερης πρόσβαση στη χρηματοδότηση. Αυτά είναι τα προβλήματα των επιχειρήσεών μας σήμερα. Σε πολλά κράτη-μέλη δεν υπάρχει πρόσβαση στη χρηματοδότηση. Έχουμε καταθέσει προτάσεις κυρίως ε, μέσω χρήσης των διαφορετικών ταμείων ως εγγυητές ε, για την ε, χρηματοδότηση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και για τα κεφάλαια κινδύνου. Και ελπίζω να προχωρήσουν αυτές οι προτάσεις. Κάναμε και συγκεκριμένες προτάσεις για να αντιμετωπίσουμε την ανεργία των νέων, μία από τις μεγαλύτερες προκρίσει που έχουμε αυτή τη στιγμή. Έχουμε κάποιες συγκεκριμένες πρωτοβουλίες και ελπίζω στο επόμενο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στις 30 Ιανουαρίου θα προχωρήσουμε σε αυτές τις προτάσεις. κοινωνική δικαιοσύνη είναι τμήμα της λύσης. Η κοινωνική δικαιοσύνη είναι σημαντική διότι θα πρέπει να υπάρχει ε, ισότιμη μεταχείριση σε όλη την κοινωνία μας. Δεν είναι αξιόπιστη η απάντησή μας χωρίς και το στοιχείο της κοινωνικής δικαιοσύνης. Ο κοινωνικός διάλογος λοιπόν είναι ζωτική σημασία και γι' αυτό ακριβώς θα συναντηθώ με τους κοινωνικούς εταίρους την επόμενη Δευτέρα στις Βρυξέλλες και ελπίζω αυτό ε, να το ακολουθήσουν ως παράδειγμα και τα κράτη-μέλη η Ευρώπη θα πρέπει να προέλθει και από εμβάθυνση της ενιαία μα αγοράς. Θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε τις δυνατότητες της πλήρω. να εγκρίνουμε μέτρα κλειδί, να έχουμε συγκεκριμένους κανόνες για τις ομοιοδετικούς διαγωνισμού, τις ηλεκτρονικές πληρωμές και τις online αγορές και επίσης θα πρέπει να δούμε και τι γίνεται ε, με ε, τις διαπραγματεύσεις για το ε, θέμα της ε, αγοράς και να, το, και να ζητήσω από τα τρία κράτη-μέλη, τη Γαλλία, τη Γερμανία και το Ηνωμένο Βασίλειο, το οποίο θεωρούν ότι το θέμα της εποπτείας το παρακολύουν, θα πρέπει να εξεύρουν σύντομα μια λύση. Δεν είναι αποδεκτό μια τόσο σημαντική πρωτοβουλία να σταματά για μια ασήμαντη διαφωνία η Ευρώπη χρειάζεται να καινοτομήσει για να αναπτυχθεί και η καινοτομία παρακολύεται από το πολύ πολύπλοκο σύστημα κανόνων που προσπαθούμε να υπερκεράσουμε εδώ και δεκαετίες. Ήγηκε η ώρα λοιπόν να γράψουμε ιστορία και να υπάρξει μία νίκη ε, για τη φιλοδοξία, για την κοινή λογική και για τους ε, Ευρωπαίους που καινοτομούν. Πολλά λοιπόν από αυτά τα οποία χρειαζόμαστε ήδη βρίσκονται στην στρατηγική ανάπτυξη τη Ευρώπη 2020. Και δεν θα μπορέσουμε να απαντήσουμε στην κρίση εάν δεν εφαρμόσουμε σοβαρά τα μέτρα αυτά. Πρέπει να υπάρχει συνέπεια σε χρονικό ε, ορίζοντα και να προσπαθήσουμε να υλοποιήσουμε τα μέτρα αυτά. Η Ευρώπη 2020 δεν είναι μια στρατηγική που μπορεί να περιμένει μέχρι το 2020. Πρέπει να δράσουμε τώρα και θα πρέπει να υπάρξει βιώσιμη ανάπτυξη. Συμφωνούμε με τη Δανία ε, για το γεγονός ότι υπάρχει προτεραιότητα για την πράσινη ανάπτυξη. Περιμένουμε η Δανική Προεδρία να ολοκληρώσει τις διαπραγματεύσεις για την ενεργειακή απόδοση την οποία παρουσιάσαμε πέρσι και να προχωρήσει και τον ενεργειακό χάρτη και τα θέματα της χαμηλής κατανάλωσης αρακά που έχουμε παρουσιάσει. Επίσης θα εξετάσει η Δανική Προεδρία και το δεύτερο ευρωπαϊκό εξάμεινο θα είναι το δεύτερο ευρωπαϊκό εξάμεινο το οποίο θα εφαρμοστεί μέσω του νέου συστήματος οικονομικής διακυβέρνησης και θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε και την εμπειρία του πρώτου εξαμήνου για να δείξουμε ότι πραγματικά μας ενδιαφέρει να μεταρρυθμίσουμε τα πράγματα και να λάβουμε πλήρως υπόψη ε, τα σοβαρά προβλήματα της οικονομίας μας. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε την ετήσια έκθεση για να υπάρχει ε, πλήρη επάρκεια χρόνου ώστε το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να εξετάσουν τα θέματα τα οποία εντοπίσαμε στην έκθεση αυτή πριν από το Εαρινό Συμβούλιο η δημοσιονομική εξυγίανση, μέτρα για την ανάπτυξη που θα προωθήσουν και την ανάπτυξη ε, πρέπει να εφαρμοστούν με αποφασιστικό τρόπο σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αξιότιμα μέλη, τα θέματα της οικονομικής ατζέντα κατά πάσα πιθανότητα θα παραμείνουν στο προσκήνιο. Θα δούμε επίσης και το νέο Δημοσιονομικό Συμβούλιο το οποίο συζητήθηκε το περασμένο Δεκέμβριο στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Είμαι πεπισμένος ότι η Ιδανική Προεδρία θα διαδραματίσει πολύ σημαντικό ρόλο και θα δράσει ως ε, προγεφύρωμα ανάμεσα στις χώρες εκτός Ευρωζώνης και εντός Ευρωζώνης. Και ελπίζουμε η Ιδανική Προεδρία να τηρήσει όχι μόνο τις αρχές της ενότητας μεταξύ όλων των κρατών μελών, αλλά να βοηθήσει και ε, στο ρόλο των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων για την ε, υλοποίηση αυτών των συμφωνιών. Υπάρχουν επίση δύο σημαντικέ συμφωνίε για την ενίσχυση τη οικονομική διακυβέρνηση στην Ευρωζώνη που παρουσίασε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τον Νοέμβριο βάσει του ε, σχετικού άρθρου τη συνθήκη και αυτά δεν περιλαμβάνονται στο λεγόμενο πακέτο των έξι οδηγιών. Επίση, θα υπάρξουν διαπραγματεύσει για το πολιετέ δημοσιονομικό πλαίσιο το οποίο θα μα βοηθήσει να έχουμε ανάπτυξη και θέσεις εργασία στην Ευρώπη τα επόμενα χρόνια. Οι συζητήσει αυτέ φυσικά θα είναι δύσκολε δεδομένων και των συνθήκων αλλά ελπίζω ότι οι προτάσει Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι ισορροπημένε αλλά και ταυτόχρονα φιλόδοξε. Και είμαι πεπισμένο ότι θα συμφωνείτε με τη φιλοδοξία τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή να δοθεί το κάθε ευρώ για να έχουμε απτά ε, χειροπιαστά αποτελέσματα για του Ευρωπαίου πολίτε. Ολοκληρώνοντα, να σα πω για τι φιλοδοξίε μα για μια ανοιχτή και ασφαλή Ευρώπη. Η Ευρωπαϊκή Ένωση πόρα απέχει από την Ευρώπη που είχαμε πριν από 10 χρόνια όταν η Δανία είχε τελευταία φορά Τότε συμμετείχα ως Πρωθυπουργός της χώρας μου στην ιστορική Ευρωπαϊκή εδώ στην Κοπενχάγη, όπου η Δανία έκανε διαπραγματεύσεις ώστε να ενταχθούν 10 νέα κράτη-μέλη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Με τον τρόπο αυτό η Δανία κατέδειξε ότι είναι διατεθειμένη να προχωρήσει με ανοιχτό τρόπο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θεωρεί ότι θα πρέπει να ενισχυθεί η φωνή της Ευρώπης και ο ρόλος της ΥΠΑ εκπροσώπου και της υπηρεσίας εξωτερικής δράσης. Επίσης, περιμένω η Ευρώπη να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στις διαπραγματεύσεις του G20 και να επιβεβαιώσει ότι έχουμε σημαντικό ρόλο για τη βιώσιμη ανάπτυξη να διαδραματίσουμε. Επίσης θέλουμε να προχωρήσει το θέμα της κοινή πολιτικής ασύλου και ε, θα ήθελα να ευχαριστήσω ιδιαίτερα για την απόφαση που ελήφθη από την Πρωθυπουργό για να σεβαστεί πλήρως την ελευθερία μετακίνησης στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ολοκληρώνοντας, κυρία Πρωθυπουργέ Τόνινγκ Σμιτ, θα ήθελα να δηλώσω ότι σε δύσκολους καιρούς όπως αυτούς είμαι πεπισμένος ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα υποφοληθεί από την προοδευτική και καινοτόμα προσέγγιση της Δανίας περισσότερο από ποτέ. Η πρόκληση είναι πάρα πολύ μεγάλη, το πρόβλημα είναι εκτεταμένο, αλλά με την κατάλληλη απάντηση και την υποστήριξη των υπολείπων θεσμικών οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης είμαι βέβαιος ότι η Δανία θα επιτύχει τους στόχους σου. Σας εύχομαι καλή επιτυχία και σας ευχαριστώ για την προσοχή σας. Ευχαριστώ πολύ κύριε Μπαρόσο. Αρχίζει τώρα η συζήτηση και ο πρώτος ομιλητής είναι ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, ο κύριος Δόλ, για πέντε λεπτά. Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κυρία Πρόεδρε του Συμβουλίου, Πρόεδρε της Επιτροπής, αγαπητοί συνάδελφοι, το να είναι κανείς πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στους τρέχοντες καιρούς δεν είναι εύκολο εγχείρημα, αλλά είμαι σίγουρος ότι μετά από την εμπειρία σας ως Ευρωβουλευτή, κυρία Πρωθυπουργέ, είσαστε οπλισμένοι με τα κατάλληλα εργαλεία για αυτό το καθήκον. Έχετε αναφέρει τέσσερι προτεραιότητε, στι οποίε έχετε βασίσει το εξάμεινό σα τη Δανική Προεδρία. Ευθύνη, δυναμισμό στην Ευρώπη, η ασφάλεια και η πρόθεση τη ζώνη του ευρώ. Εγώ με τι απόψει σα. Όπω ξέρουμε όλοι, <clears throat> οι προεδρίε δεν μπορούν να διαλέξουν την ημερησία διάταξή του. Είναι η πολιτική πραγματικότητα η οποία είναι το οδηγό νήμα κάθε προεδρία. Γι' αυτό ζητώ από την ιδανική Προεδρία να μην περιοριστεί να είναι μονάχα μια τεχνικού χαρακτήρα προεδρία, αλλά να είναι μια πολιτική προεδρία, λαμβάνοντα υπόψη την ευρύτητα των προβλημάτων που έχουμε ενώπιό μα και πρέπει να αντιμετωπίσουμε. Για τον λόγο αυτό σα ζητώ επίση και ζητώ και από την ιδανική Προεδρία να συνεργαστεί στενά με το Κοινοβούλιο που γνωρίζετε τόσο καλά, αλλά που ορισμένες από τις κυβερνήσει θέλουν να παίξει το ρόλο απλώς ενός διαδικαστικού σώματος. Αυτό δεν το δεχόμαστε όλοι. Υποστηρίζουμε με την ταχύτητα της νομοθεσίας και μας διδάσκουν οι αγορές ή μας υποχρεώνουν περισσότερο τον, περισσότερο των τα πρώτα τις πρόσφατες μέρες να εργαζόμαστε με ταχύτητα. Αλλά πρέπει συγχρόνως να εξασφαλίσουμε την καλή λειτουργία της δημοκρατίας και την διαφάνεια. Είμαι σίγουρος κύριε Πρόεδρε ότι η Προεδρία σας θα βρει ένα σωστό, μια σωστή θέση δίπλα στο Κοινοβούλιο και την Κομισιόν και σας ζητώ να αποδεθείτε στην πολιτική. Γιατί <clears throat> πρέπει να υπάρξει πραγματικά μια δράση από τους πολιτικούς άνδρες και γυναίκες της Ευρώπης να είναι όχι μονάχα δεσμευμένοι στην ιδέα της Ευρώπης, αλλά να είναι ορατοί και ακουστοί. Έχει ξεκινήσει η διαπραγμάτευση της νέας διακυβερνητικής συνθήκης. Εμείς από το Κοινοβούλιο περιμένουμε ακόμα να έχουμε μια συζήτηση για τα θέματα αυτά. Ελπίζουμε ότι θα εμπλακούμε πλήρως στη διαπραγμάτευση αυτής της συνθήκης και ελπίζουμε ότι δύο βασικές αρχές θα γίνουν σεβαστές από το Συμβούλιο. Η αρχή τη ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης στα θέματα του προπολογισμού και τα δημοσιονομικά, αλλά επίσης και σε πολιτικό επίπεδο και στο επίπεδο της διατήρησης της κοινοτική της ενωσιακή μεθόδου. Επιπλέον θέλω να σα υπενθυμίσω ότι η ομάδα του ΕΛΚ θα σα είναι ευγνώμων αν μπορέσετε να θέσετε σε σωστή τροχιά τις πρώτες συζητήσεις για τι δημοσιονομικέ προοπτικές τη Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν είναι εύκολο το θέμα αυτό, χρειάζεται τόλμη από εσά. Οι μεταρρυθμίσει που θέλετε να επιφέρετε στα δημόσια οικονομικά και για να επανέλθει η οικονομική ανάκαμψη και ανάπτυξη είναι η πρώτη σα προτεραιότητα. Δεν πρέπει όμω να ξεχάσουμε και την σημαντική συζήτηση για τα δημοσιονομικά της Ευρώπης στη χρονική περίοδο 2014-2020. Κάθε ευρώ λοιπόν το οποίο χρησιμοποιείται από εσά και την Κομισιόν είναι ένα πραγματικό ευρώ. Και από κάθε ευρώ το οποίο δίνεται στις χώρες που έχουν μεγάλα ελλείμματα είναι ένα ευρώ το οποίο θα πρέπει να οδηγήσει και στην ανάπτυξη. Αν μπορέσει η Ιδανική Προεδρία να ξεκινήσει χωρίς ταμπού και χωρίς ε, προκαταλήψεις στη συζήτηση για τους ίδιους πόρους, αν μπορέσει να πείσει τα κράτη-μέλη ότι το να δαπανούνται χρήματα σε ευρωπαϊκό επίπεδο σε μεγάλα οριζόντια σχέδικα είναι καλύτερο παρά να κατακαιρματίζονται αυτά τα ποσά και να δαπανώνται μονάχα σε εθνικό επίπεδο, τότε θα έχετε την πλήρη αναγνώριση αυτού του Κοινοβουλίου. Κυρία Πρόεδρε, είναι απαραίτητη η αποτελεσματικότητα και το θάρρο των Προεδριών που πολλές φορές βλέπουμε περισσότερο στις λεγόμενες μικρές Προεδρίες. Είναι λοιπόν η ευκαιρία για εσά, όπως και η Πολωνία πριν από εσά, να δείξετε φιλοδοξία και ακόμα και σε θέματα όπως είναι η νομισματική πολιτική θα πρέπει να δείξετε τόλμη στις προτάσεις σας και <clears throat> μαζί με το Κοινοβούλιο να πείσετε τα κράτη-μέλη ότι η λύση των προβλημάτων της Ευρώπης περνάει από περισσότερη Ευρώπη, περισσότερη σύγκριση και, σύγκληση συγγνώμη, και αυτό θα υποστηριχθεί πολύ περισσότερο σε αυτή την περίπτωση από τους συμπολίτε μας. Σας εύχομαι καλή τύχη το επόμενο εξάμεινο. Ευχαριστώ πολύ, ο Πρόεδρος. Κύριε Ντόλ για την Σοσιαλιστική και Δημοκρατική Ομάδα έχει το λόγο ο κύριος Φόμποντα, τον οποίο συγχαίρω και για την εκλογή του ως επικεφαλής της Σοσιαλιστικής Ομάδας του Ευρωπαϊκό κοινοβουλίου. Για 5,5 λεπτά έχει το λόγο ο κύριος Φόμποντα. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Και εγώ μπορώ να σας ευχαριστήσω και να σας συγχαρώ για την εκλογή σας. Θέλω λοιπόν να σας ευχαριστήσω και για την γενεοδορία σας σε σχέση με τον χρόνο αγόρευσης. Κυρία Πρόεδρε του Συμβουλίου, κύριε Πρόεδρε της Επιτροπής, συζητούμε για την Ευρώπη σε μια δύσκολη χρονική στιγμή. Η Ευρώπη πρέπει να παίξει ένα ρόλο σε ένα πλαίσιο όπου αυτοί οι οποίοι κινούν τα νήματα είναι οι παίκτες στις χρηματαγορές που δεν είναι παρόντες εδώ σήμερα. Πρέπει λοιπόν να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα αυτά στα οποία δεν είναι άμυρες και ευθύνη οι φορείς πιστοληπτικής αξιολόγησης. Πρέπει να ξεπεράσουμε λοιπόν αυτές τις αδυναμίες της Ευρώπης. Να βρούμε λύσεις όπως το παρελθόν που πολλές φορές ήταν πάρα πολύ δύσκολες. Το δείχνουν οι φορείς πιστοληπτικής αξιολόγησης ότι αν δεν υπάρχει μια κοινή δράση στην Ευρώπη, εμείς θα κινήσουμε τα νήματα, λένε αυτοί οι φορείς. Ελήψη Ευρώπης όπως ανέφερε και η πρόεδρος του Συμβουλίου, είναι ένα θέμα όχι μόνο των αγορών, αλλά και των ανθρώπων. Θα πρέπει να βγούμε λοιπόν από μια σαφή, από μια πολιτική μόνο λιτότητας. Και εκεί είναι σαφής οι φορείς πιστοληπτικής αξιολόγησης που είπαν ότι με μια τέτοια μονομερή πολιτική αυστηρότητας δεν θα μπορέσουν να ξεπεραστούν τα προβλήματα των προϋπολογισμών. Το τόνισε και, το, και η Financial Times όταν είπαν ότι η δημοσιονομική συνθήκη που είναι ε, το κυριότερο θέμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης αυτή τη στιγμή είναι άσχετο προς την πραγματικότητα. Είναι μια ασήμαντη λεπτομέρεια. Πρέπει λοιπόν να προχωρήσουμε μεν σε σχέση με το θέμα αυτό, αλλά θα πρέπει να λάβουμε υπόψη τι γίνεται αυτή τη στιγμή στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι σαφές ότι αυτή η πολιτική λιτότητα είναι μια αντικοινωνική πολιτική. Δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να έχουμε εξοικονόμηση, αλλά αυτό δεν πρέπει να γίνεται σε βάρος των πολιτών και των ασθενεστέρων. Θα ήθελα να κάνω μια έκκληση σε όλους. Να ξαναβρούμε το σωστό δρόμο, ο οποίος θα εξασφαλίσει το κοινωνικό κράτος στην Ευρώπη. Γιατί χωρίς κοινωνικό κράτος δεν θα μπορέσουμε να ξεπεράσουμε τα προβλήματα των προϋπολογισμών. θα πρέπει να μην αμφισβητήσουμε τη σημασία του κοινωνικού κράτους γιατί αυτό αλλιώς θα μας οδηγήσει σε αναταραχές, σε περιστολή των ε, δικαιωμάτων των πολιτών. Είδαμε αυτά τα οποία έγιναν στο Βουκουρέστι και σε άλλες πόλεις της Ρουμανίας ήδη σε, λόγω αυτών των προβλημάτων. Έχουμε ακούσει για τους στόχους της Λισαβόνας που είχαμε θέσει ότι θα έπρεπε να γίνουμε η πιο ανταγωνιστική περιοχή του κόσμου χάρη στην, χάρη στην ε, πληροφορία και τη γνώση και την κοινωνία της πληροφορίας. Μιλήσατε επίσης για τις μελλοντικέ γενναίες, κυρία Πρόεδρε του Συμβουλίου. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Είπατε πολύ σωστά στο πρόγραμμά σας ότι η Ευρώπη θα πρέπει να δημιουργήσει τη δυνατότητα θέσεων εργασίας, να ξεπεράσουμε την ανεργία. Προφανώς και η δική μου ομάδα θέλει να δώσει έμφαση στην Ευρώπη της εργασίας. Αυτό όμως μπορεί να γίνει μονάχα και εδώ θέλω να είμαι απόλυτα σαφής όταν τονίσουμε την ανάγκη να υπάρχουν και πράσινες θέσει εργασία και συνδέσουμε απόλυτα την οικολογία με τις πολιτικές που ακολουθούμε. Όχι να τις θέσουμε σε αντιπαράθεση. Πρέπει να αγωνιστούμε όλοι για να υπάρχουν νέε θέσει εργασία, ενώ συγχρόνω προστατεύουμε το περιβάλλον και έχουμε μια πορεία ανάπτυξη η οποία να είναι πραγματικά αηφόρο. Τότε θα σα υποστηρίξουμε απόλυτα, κυρία Πρόεδρε του Συμβουλίου, γιατί και η ενεργειακή απόδοση είναι κάτι το οποίο μα ενδιαφέρει ιδιαίτερα. Θέλουμε να έχουμε μια αποδοτική χρήση τη ενέργεια. Έχουμε πολύ καλά παραδείγματα τα οποία πρέπει να τα μιμηθούμε. Και αυτό που είναι απαραίτητο είναι να μπορέσουμε να ανακτήσουμε την υπερηφάνεια στο ευρωπαϊκό εγχείρημα. Όταν βλέπουμε τους Αμερικανούς, τους Κινέζους, έχουν και αυτοί αντιμετωπίσει πολλά προβλήματα στο παρελθόν, αλλά έχουν ξεπεράσει κάποια από αυτά. Ελπίζω ότι μετά τη Δανική Προεδρία θα μπορούμε να πούμε το ίδιο και για την Ευρώπη. Δεν θέλω λοιπόν να ξεπεράσω την, ε, το χρόνο μου <clears throat> και θα ήθελα να περιοριστώ μονάχα σε μια σύντομη παρατήρηση. Να πω ότι σαν πολιτική ομάδα είχαμε μια πάρα πολύ θετική αντιμετώπιση στην ε, διαδικασία ε, εκλογής του νέου Προέδρου της Σοσιαλιστικής Ομάδος. Και θέλω να ευχαριστήσω και τους αντιποψηφίους μου, την κυρία Τροτμάν και τον κύριο Χιούς. Είναι σημαντικό λοιπόν αυτό και για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και για την Κομισιόν και το το Συμβούλιο. Έχουμε όλοι μας μια νέα, μια διαφορετική εικόνα της Ευρώπης, μιας Ευρώπης με αλληλεγγύη, μιας Ευρώπης η οποία έχει κοινωνικό χαρακτήρα. Ε, έχουμε διαφορές απόψεις μαζί σας με το Συμβούλιο και την Κομισιόν ορισμένε φορές, αλλά όλα αυτά τα θέματα θα πρέπει να είναι αντικείμενο συζήτησης. Θέλω λοιπόν να τονίσω τη σημασία να υπάρχει διάλογο σε αυτό το Κοινοβούλιο και θέλω να ευχαριστήσω και τον Πρόεδρο για την υπομονή που έδειξε με τον χρόνο αγόρευσης. Ευχαριστώ πολύ. Τώρα για την φιλελεύθερη και δημοκρατική ομάδα έχει το λόγο ο κύριο Γκίφερ Χόφστατ. Ε, ευχαριστώ πρόεδρε. Κύριε Πρωθυπουργέ, κυρία Πρωθυπουργέ, μία προτεραιότητα έχετε. Να βρείτε το δρόμο να βγούμε από τις δύο κρίσεις που ζούμε. Την ευρωκρίση και την κρίση των ευρωπαϊκών αξιών. Κάτι σαφές, που είναι σαφές είναι ότι τα μέτρα που έχουν ληφθεί τα τελευταία δύο χρόνια δεν απέδωσαν. Σε όλες τις διμερείς συναντήσεις Μέρκελ και Σαρκοζή τίποτα δεν απέδωσε. Για 24 ώρες φαίνεται ότι κάτι αντιμετωπίζεται και μετά ξαναρχίζουν τα πράγματα όπως πριν. Οι κερδοσκόποι έχουν επιτεθεί σε όλες τις ευρωπαϊκές κυβερνήσεις. Δεν είμαι και εγώ υπέρμαχος των ε, οργανισμών αξιολόγησης, αλλά δεν αξίζει τον κόπο να παραπενούμεθα για, αυτές, για αυτούς. Ας διαβάσουμε καλύτερα τι μας λένε και τι μηνύματα μας δίνουν. Αυτό που μας λένε είναι σωστό. Απογοητεύτηκα από ο κύριος Μπαρνιέ και άλλοι παραπονέθηκαν, γιατί άμα διαβάσει κανείς τι λέει η Standard και Πούρ είναι αλήθεια αυτό που λένε ότι υπάρχει δηλαδή έλλειψη πολιτικού θάρρους και ενότητας στην Ευρώπη και λένε και αυτοί ότι δεν είναι μόνο δημοσιονομική κρίση αλλά και κρίση εμπορικής έλλειψης ισορροπίας έλλειψης ε, στα ισοζύγια ορισμένες χώρες μειώνουν τις δαπάνες τους για να μπορέσουν και αυτές να αναπτυχθούν αλλά λένε στάνταρτ και πούρς ότι χρειάζεται ανάπτυξη. Βλέπω ότι μερικοί χειροκροτούν του στάνταρτ και πούρ. Ο λένε λοιπόν ότι μόνο μία βιώσιμη λύση θα μπορεί να πρέπει να βρεθεί η οποία θα είναι αναπτυξιακή και αυτή δεν προτείνεται από κανέναν. Χρειαζόμαστε σταθερότητα, ό,τι πως θέλετε πέστε το, αλλά και η γερμανική πρόταση του Ταμείου Ανάνυψης δεν θα επιφέρει αποτελέσματα. Δεν είναι δικές μου απόψεις αυτές. Είναι το σημερινό μήνυμα και του Πρωθυπουργού της Ιταλίας, του Financial Times. Λέει, εγώ δεν παραπονούμε για την υποβάθμιση, γιατί το πρόβλημα είναι ότι συνεχίζεται η πολιτική αδυναμία της Ευρώπης. Ο Μάριο Μόντι το λέει σήμερα στους Financial Times. Και τι άλλο λέει. Χρειάζεται απλώς η κυρία Μέρκελ να μου χαϊδέψει τον νόμο για να με παρηγορήσει. Πρέπει να δεχτεί τα ευρωομόλογα. Και έχει δίκιο, δεν υπάρχει βιώσιμη λύση. Αλλιώς με επιτόκια 6 και 7%. Ο μόνος τρόπος να βγούμε από την κρίση είναι να ληφθούν μεν αυτά τα μέτρα με χαμηλότερα επιτόκια, όχι 6-7%. Αλλιώς ζητούμε από τον κύριο Μόντι κάτι που δεν μπορεί να το πραγματοποιήσει του λέμε μπράβο μπράβο παίρνεις μέτρα λιτότητας αλλά δεν μπορούν αυτά να εφαρμοστούν καν με τέτοια επιτόκια και δεύτερον κυρία Πρωθυπουργέ υπάρχει ένα δεύτερο πρόβλημα μια δεύτερη κρίση των αξιών δέστε τι έγινε σήμερα στη Ρουμανία η Κομισιόν είπε, έκανε προσφυγές και ελπίζω και εμείς εδώ στο Κοινοβούλιο με πλειοψηφία να καταφέρουμε να εφαρμόσουμε το άρθρο 7 να προσφύγουμε δηλαδή. Και ερωτώ τον κύριο Πιτέλα, τον οποίο συγχαίρω για την εκλογή του, που μου έδωσε περισσότερο χρόνο γι' αυτό τον συγχαίρω. Μα είστε Ιταλός, το κάνουν αυτό στην Ιταλία. Δίνουν ο ένας το χρόνο στον άλλον. Λοιπόν, κυρία Πρωθυπουργέ, προσφεύγει η Κομισιόν και εμείς αρχίσουμε μια διαδικασία με βάση το άρθρο 7 αλλά το Συμβούλιο τι θα κάνει, θα το συζητήσει την επόμενη του συνεδρίαση γιατί νομίζω θα ήταν λάθος να μην το κάνει. Γιατί το θέμα της Ευρώπης δεν είναι μόνο τα λεφτά αλλά και οι ελευθερίες και οι αξίες. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Φερχόφστατ. Σας ευχαριστώ όλους. Καλημέρα σας. Θα ήθελα να ρωτήσω τον κύριο Φερχόφστατ αν μπορεί να απαντήσει σε μια ερώτηση που θέλει να του διατυπώσει ο κύριος Γκαργκάνη, αν δεν κάνω λάθο. Α, μετά, στο κάτσε διά, να μιλήσετε. Ε, νόμιζα ότι ζητήσετε μπλε κάρτα. Τέλος πάντων, ωραία. Να προχωρήσουμε με τη συζήτηση. Η κυρία Ρεμπέκα Χάρμ για τέσσερα λεπτά έχει το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κυρία Πρόεδρε του Συμβουλίου, είναι μια μεγάλη τιμή για μένα που μπορώ να σας καλωσορίσω εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και γνωρίζετε πολύ καλά ότι η πολιτική μου ομάδα υποστηρίζει την κόκκινη-κόκκινη πράσινη κυβέρνηση στην ε, Δανία και έχει ιδιαίτερες προσδοκίες από εσά, όχι μόνο λόγω της πολιτικής σας προέλευσης και του τόσο ενδιαφέροντος νέου σχήματος που κυβερνά τώρα την ε, ε, Δανία, αλλά διότι πιστεύω ότι με την σκανδιναβική σας ευρωστία μπορείτε να προτείνετε μια νέα κατεύθυνση για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και νομίζω ότι η γοητευτική σας νυφαλιότητα στην πολιτική που εκπορεύεται από την Κοπενχάγη θα μπορέσει να αποτελέσει και ένα τρόπο να πείσετε την θηλυκή ομόλογό σας στη Γερμανία να ακολουθήσει μια κάπως διαφορετική πολιτική. Αυτό περιμένουμε από εσά. Περιμένουμε ότι την ε, συνθήκη αυτή που συζητείτε μετά από την τελευταία διάσκεψη κορυφής να την αντιμετωπίσετε με κριτικό πνεύμα. Γιατί αυτή η συνθήκη δεν πρέπει να είναι μονάχα μία τεχνική λύση αλλά και μία ενθάρρυνση για την Ευρωπαϊκή Ένωση να συμπεριλάβει και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τα Εθνικά Κοινοβούλια και να τα εμπλέξει περισσότερο και όχι να συνεχίσει σε αυτή την απαράδεκτη μέχρι τώρα οδό. Πιστεύω ότι η διάσκεψη κορυφής για το ευρώ που μέχρι τώρα ήταν άτυπη και στο μέλλον θα είναι επίσημη και εκεί θα πρέπει η Δανία να προσπαθήσει να εξασφαλίσει την καλύτερη ισορροπία δυνάμεων στο Συμβούλιο. Όλα αυτά λοιπόν τα οποία είναι θέματα δύσκολα σε τεχνικό επίπεδο δεν πρέπει να αποκρύψουν τις δημοκρατικές α, ανησυχίες οι οποίες έχουν πολύ μεγάλη σημασία για το μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σε ό,τι αφορά το περιεχόμενο αυτό έχει επικριθεί από όλους τους προλαλήσαντες ομιλητές η συνθήκη αυτή γιατί δίνει έμφαση μονάχα στη σταθερότητα και τη λιτότητα και αυτά δεν αντιμετωπίσαν την κρίση, έχουν μάλλον οξύνει ακόμα περισσότερο την κρίση. Και μπορώ να σας υποσχεθώ ότι σε κάθε ολομέλεια θα βλέπετε να θα είστε υποχρεωμένοι να καταλαβαίνετε και να διαπιστώνετε ότι τα πράγματα είναι πολύ χειρότερα από την προηγούμενη. Ε, η Παγκόσμια Τράπεζα τονίζει τόνισε πρόσφατα ότι η Ευρώπη αυτή τη στιγμή πέφτει όλο και βαθύτερα στην κρίση και τραβάει όλο τον πλανήτη μαζί της. Στο πρόγραμμά σας, το πρόγραμμα της Ιτανικής Προεδρίας, έχετε κάποια στοιχεία τα οποία είναι υπόσχεση μιας διαφορετικής πορείας. Αλλά θα πρέπει να μην περιμένετε μέχρι τη μέση ή το τέλος του εξαμήνου σας για να μπορέσετε να προωθήσετε αυτό το πρόγραμμα επενδύσεως για την ανάκαμψη της οικονομίας. Οι ιδέες σας για την προστασία του περιβάλλοντος που νομίζω ότι έχουν προετοιμαστεί τα μάση από την Κόνι Χέντεγκα, την αρμόδια επίτροπο. Όλα αυτά μπορούν να είναι η λοκομοτίβα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης. Δεν πρέπει να χάσετε λοιπόν άλλο χρόνο για να τα εφαρμόσετε όλα αυτά. Για την δημιουργία επίσης ενός πλέγματος ρύθμισης των χρηματαγορών. Και αυτό αναφέρθηκε από πολλούς ομιλητές. Εγώ συμφωνώ να υπάρξει η υποστήριξη του Ταμείου ε, Ανακύλησης και τα, την χρήση των ευρωπαϊκών ομολόγων. Αλλά να πω και κάτι για το ρόλο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας σε αυτή την κρίση, γιατί και αυτό αποτελεί, όπως και στο παρελθόν, ένα μεγάλο πρόβλημα. Έχουμε ένα κοινό νόμισμα το οποίο θέλουμε να υποστηρίξουμε, αλλά δεν έχουμε προχωρήσει προς την κατεύθυνση του να έχουμε <clears throat> μια κεντρική τράπεζα η οποία λειτουργεί πραγματικά ενωσιακή και η οποία θα πρέπει να έχει την απαραίτητη εξουσιοδότηση από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Σταθερότητος. Αναφέρθηκε από πολλούς ομιλητές το πρόβλημα των ε, φορέων πιστοληπτικής αξιολόγησης και δεν έχουν καταλάβει ακόμα τα κράτη-μέλη ποια είναι τα αποτελέσματα και οι απόρριες αυτών των υποβαθμίσεων. Θα ήθελα λοιπόν αγαπητοί πρώην συνάδελφε, ε, πρόεδρε του Συμβουλίου, θα θέλαμε να σας ζητήσουμε να κάνετε τα πράγματα καλύτερα από τους προκατόχους σας. Να δράσετε τώρα, να πάρετε τα απαραίτητα βήματα, να αντανακλαστεί και η πολιτική σας πεποίθηση στο Συμβούλιο αυτά που θα συζητήσουμε το απόγευμα είναι πάρα πολύ σημαντικά. Σαν παράδειγμα, πώς η Κομισιόν και το Συμβούλιο έχουν αφήσει ένα πρόβλημα να χρονίζει και ουσιαστικά τώρα πρέπει να πληρώσουμε την ύφη για αυτά τα οποία έγιναν στην Ουγγαρία. Τα επίχειρα μιας ε, αβελτηρίας του Συμβουλίου και της Κομισιόν για να αντιμετωπιστεί αυτή η κρίση. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας. Ευχαριστώ κυρία Χάρμς. Ο λόγος τώρα στο Μάρτιν Κάλαναν για τρία λεπτά. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Συγγνώμη, συγγνώμη, διακόπτει ο Πρόεδρος. Κύριε Κάλαναν, συγγνώμη σας διακόπτω. Κάποιος έχει ζητήσει να χρησιμοποιήσει μπλε κάρτα. Μπορεί η κυρία Χάρμς να απαντήσει. Παρακαλώ, κυρία Μορβόη, ευχαριστώ. Αν δεν κάνω λάθος, κυρία Χάρμς, είπατε ότι η Ουγγαρία είναι αυτή η οποία πρέπει να κατηγορήσουμε για όλα τα κακά τα οποία μας αναφέρατε στην ομιλία σας. Η Ουγγαρία έχει το φταίξιμο και για την κρίση και για όλα τα υπόλοιπα. Και πώς συσχετίζεται το ουγγρικό ζήτημα με όλα όσα είπατε. Σας ευχαριστώ πολύ ist ein Land mit erheblichen wirtschaftlichen Problemen. Ναι. Ναι. Υπάρχουν πραγματικά σοβαρά οικονομικά προβλήματα που αντιμετωπίζει η Ουγγαρία και η κυβέρνηση του Βίκτορ Ορμπάν δεν βρήκε καμία διέξοδο από τα προβλήματα αυτά. Αντί του να βρει μια λύση, χρησιμοποίησε το σοβινιστικό εθνικιστικό χαρτί στην Ουγγαρία, ώστε να μπορέσει να καλύψει την αδυναμία της δικής του πολιτικής στην Ουγγαρία. Εγώ υποστηρίζω ότι πρέπει μαζί με τους Ούγγρους, όπως και με οποιοδήποτε άλλο κράτος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να αντιμετωπίσουμε με αλληλεγγύη τα κοινά οικονομικά προβλήματα. Αλλά η αλληλεγγύη δεν είναι μια αξία την οποία μπορεί να χρησιμοποιεί κανείς όποτε θέλει και αλλιώς να αποκλείει άλλες αξίες. Η Ευρωπαϊκή Ένωση βασίζεται στην αλληλεγγύη αλλά και με ένα πλέγμα άλλων αξιών και αυτό δεν πρέπει να το ξεχάσει η κυβέρνηση του Βίκτορ Ορμπάν. Σας ευχαριστώ. Να ξαναδώσουμε λοιπόν τώρα το λόγο στον κύριο Κάλαναν για τρία λεπτά. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Καταρχάς να καλωσορίσω την κυρία Τόρνινγκ Σμιθ ε, σήμερα στην έδρα και να σας ε, συγχαρώ διότι πλέον ένα μέλος ε, της οικογένειάς σας γίνεται πλέον πρωθυπουργός. Κάποιο τα κατάφερε, θα χαρεί το Ηνωμένο Βασίλειο. Η Δανία είναι ιστορικό σύμμαχο και η Δανία και με το προσωπικό της υπηρέτησε με τη χώρα μου και με Γάλλους επικόους ε, για να βοηθήσει ε, τη Λιβύη και σας ευχαριστώ γι' αυτό. Και χαίρομαι που η Δανία ανέλαβε την Προεδρία σε μια τόσο κρίσιμη στιγμή όταν βρισκόμαστε στο χείλος της πολιτικής και της οικονομικής καταστροφής. Και ελπίζω η Δανική Προεδρία να μπορέσει να μιλήσει με απλά λόγια. Πολλές φορές λέμε ότι οι πιο θεραλές πράξεις, ε, οι πιο πράξεις στην πολιτική είναι να λέμε με την αλήθεια. Και νομίζω ότι η Δανική Προεδρία τα, έκανε, ε, τα πήγε καλά μέχρι τώρα με την ειλικρινή αξιολόγηση τη οικονομική ε, καταστροφή και το τι στήχησε αυτό στην Ευρώπη. Και ελπίζω να πείσει όλου του ηγείτε τη Ευρωπαϊκή Ένωση ότι πλέον έφτασε το πλήρωμα του χρόνου να αντιμετωπίσουν την αλήθεια κατά πρόσωπο και να δούνε όλε τις αδυναμίε. Διότι το τελευταίο Συμβούλιο ήταν μια πραγματικά χαμένη ευκαιρία. Αντί να αντιμετωπίσουν την πραγματικότητα και να αντιμετωπίσουν τα προβλήματα, ξεκίνησαν ένα έναν νέο γύρο ενδοσκόπησης και ομφαλοσκόπησης. Δεν θα πρέπει να ξεχνούμε ότι βρισκόμαστε εν μέσω όχι μίας αλλά δύο πολύ μεγάλων κρίσεων. Βεβαίως η, Ευρωπαϊκή, η Ευρωζώνη είναι το πιο άμεσο πρόβλημα αλλά δεν θα πρέπει να ξεχνάμε το γεγονός ότι αντιμετωπίζουμε μια θεμελιώδη πρόκληση για την οικονομική μας κατάσταση. Χάνουμε την ανταγωνιστικότητα στην παγκόσμια αγορά, ε, αντιμετωπίζουμε ε, απώλειες από πιο δυναμικές περιοχές ανά τον κόσμο, χάνουμε τη δυνατότητα δυνατότητα ε, να κάνουμε τις κατάλληλες νομοθεσίες και έχουμε ρυθμίσεις που παρακολύουν την καινοτομία. Χρειαζόμαστε μια ανάπτυξη λοιπόν η οποία θα μας βοηθήσει να δημιουργήσουμε νέες θέσεις εργασίας και να βοηθήσουμε τις επιχειρήσεις. Θα πρέπει να δημιουργήσουμε τις κατάλληλες μεταρρυθμίσεις και να αναπτύξουμε την ενιαία αγορά και θα πρέπει να υποστηρίξουμε λοιπόν κάποιες από τις βασικές προτεραιότητες της Ιδανικής Προεδρίας. Για το πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο συμφωνούμε ότι θα πρέπει να το εξετάσουμε ε, μέσω της εξυγίασης των δημοσίων οικονομικών και θα πρέπει να εξετάσουμε το μέλλον και όχι το παρελθόν. Να υπάρχει κατάλληλη αποτελεσματικότητα και όλα αυτά τα οποία είπατε για αυτό το θέμα είναι ευπρόσδεκτα. Όλα τα κράτη-μέλη θα πρέπει να δουν με αντίστοιχο ρεαλιστικό τρόπο τον ευρωπαϊκό προπολογισμό. Θέλουμε να παγώσει ο προπολογισμό και να επικεντρωθούμε στην κατάλληλη χρήση των, ε, ε, των κονδυλίων που έχουμε στη διάθεσή μα αυτή τη στιγμή. Θα πρέπει επίσης ε, ε, να συμφωνήσουμε και με αυτό που είπε ο Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να αναζωογονήσουμε την Ευρωπαϊκή Ένωση διότι είναι μια ανοιχτή περιοχή για τις επενδύσεις. Το να είμαστε οικονομικά ανοιχτά σημαίνει ότι θα αυξηθεί και η ανάπτυξη και η, ε, θα πατάξουμε την ανεργία. Θα πρέπει λοιπόν να χρησιμοποιήσουμε ορολογία 21ου αιώνα για να λύσουμε τα προβλήματα του 20ου αιώνα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναφέρεται σε περισσότερη νομοθεσία, σε υπεύθυνη οικονομία και σε οικονομία οικονομική ε, στασιμότητα. Δεν θα πρέπει λοιπόν να λησμονούμε ότι οποιασδήποτε πλεερητέρω νομοθεσία έχει το κόστος του, το οποίο κόστο είτε το πληρώνουν οι καταναλωτέ όταν αγοράζουν αγαθά, είτε από τι υπηρεσίε που ε, ε, πληρώνουν ή από του εργαζόμενου που χάνουν τις θέσει εργασία του από ανθρώπου που έρχονται ε, από άλλε χώρε. Δεν θα πρέπει λοιπόν να κρυφτούμε πίσω από τις ε, πρωτοβουλίε, θα πρέπει να λάβουμε κατάλληλες δράσεις για τι εξωτερικέ σχέσει και τι εσωτερικέ υποθέσει. Θα πρέπει επίσης να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε ε, αυτές τις επικίνδυνες προτάσεις που γίνονται για τους φόρους, ε, για τις ε, συναλλαγές και θα πρέπει να προχωρήσουμε όλα τα θέματα. Καλωσορίζουμε λοιπόν τη Δανική Προεδρία και την ευχαριστούμε για τη διάθεση που θα επιδείξει. Ευχαριστούμε. Ο λόγος τώρα για τρία λεπτά στον κύριο Σόντεγκαρντ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Θα ήθελα να ξεκινήσω συγχαίροντας την, ε, την ε, Δανική Προεδρία και την Δανική Κυβέρνηση. Να σας συγχαρώ γιατί περάσατε 100 ημέρες στην εξουσία ως ε, νέα δανική κυβέρνηση μετά τις εκλογές του Σεπτέμβριο. Η Γέννη Τόλι Σμιτ και η συμμαχοί της έθεσαν ένα σαφές ερώτημα το οποίο κλήθηκε να απαντήσει ο λαός της Δανίας. Θα πρέπει να επενδύσουμε για να εξάλλουμε τις κρίσεις ή θα πρέπει να κάνουμε οικονομίες για να βγούμε από την κρίση, να λύσουμε την κρίση δημιουργώντας θέσεις εργασίας ή ανεργία. Ο λαός της Δανίας απάντησε εκλέγοντας τη χέρι Σμιτ στη θέση της Πρωθυπουργίας. Το θέμα όμως και το ερώτημα που τέθηκε κατά την προεκλογική εκστρατεία στη Δανία είναι ακόμα πιο απαραίτητο και σχετικό, αν θέλετε, για την ευρωπαϊκή οικογένεια. Γιατί η Ευρωπαϊκή Ένωση διανύει την πιο βαθιά κρίση που έχει περάσει ποτέ. Πάνω από 10% των πολιτών της Ευρώπης είναι άνεργοι. 5 εκατομμύρια στην Ισπανία και μόνο. πληθυσμό μεγαλύτερο από την ε, Δανία. Δύο τρίτα των ευρωπαϊκών κρατών έχουν 30, 40% ενεργεία στους νέους, 40% στην Ελλάδα, 50% ακόμα στην Ισπανία μεταξύ των νέων. Το πρόγραμμα για την Ιδανική Προεδρία φαίνεται ότι έχει γραφτεί από το Μερκοζή. Μας απογοητεύει αυτό. Και χάθηκε η ιδέα της επένδυσης για να ξεπεράσουμε την κρίση. Τώρα μόνο περικοπές ε, βλέπουμε. Οικονομία για να λύσουμε την κρίση. Μα πιστεύει κανείς ότι με την λιτότητα μπορούμε να βγούμε από την κρίση. Η Ευρωπαϊκή Ένωση το δοκίμασε στην Ελλάδα. Δεν το πέτυχε. Το ξαναπροσπάθησε πάλι η Ευρωπαϊκή Ένωση στην Ελλάδα και πάλι χωρίς επιτυχία και τώρα τρίτη φορά προσπαθούν να το πετύχουν στην Ελλάδα και πάλι δεν υπάρχουν ενδείξεις ότι πρόκειται να πετύχει. Το πρόγραμμα της Δανικής Προεδρίας έχει τον τίτλο «Η Ευρώπη δουλεύει, Europe at Work». Αλλά η πολιτική που βλέπουμε ότι μας παρουσιάζεται θα οδηγήσει σε περαιτέρω ανεργία. Η ομάδα μας θεωρεί ότι κινούμαστε προς τη λάθος κατεύθυνση. Άρα θα ήθελα να κλείσω λέγοντας προς την Δανική Προεδρία ότι οι λαοί της Ευρώπης δεν χρειάζονται πιο πολλές περικοπές που θα υπαγορεύονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν, χρειάζομαι, δεν χρειαζόμαστε δημοσιονομικές επιταγές για να μειώσουν τις υπηρεσίες μας, για να περικόψουν τους μισθού μας. Όχι, χρειαζόμαστε θέσεις εργασίας, χρειαζόμαστε βελτίωση της ευημερίας και η Ιδανική Προεδρία έχει έξι μήνε στη διάθεσή τη για να μα καταδείξει ότι αποτελεί τμήμα τη Λύση και όχι τμήμα του προβλήματο. Σα ευχαριστώ πολύ. Ε, ευχαριστώ συνάδελφε. Ο κύριο Μέσσερ Σμιτ για δύο λεπτά. Ε, ευχαριστώ πολύ πρόεδρε. Ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρον ε, εδώ και 30 λεπτά να είμαι μάρτυρας μιας love story μίας ιστορίας αγάπης. όπου διαπιστώνουμε ότι μετά από μία κατάρτιση στο Ευρωπαϊκό Κολέγιο της Μπρούζ ε, η Πρωθυπουργό, ε, βάσει μιας απάτης έγινε Πρωθυπουργό, γιατί τελικά κανένας εκλογέας δεν ψήφισε υπέρ αυτή. Πολλοί δανείοι εκλογής ε, θεωρούν ε, σήμερα ότι παρασύρθηκαν να υπερψηφίσουν την Τόνε Σμιτ αλλά αυτό δεν συνέβη, δεν έπρεπε να γίνει. Στην Ελλάδα και στην Ιταλία χρειάστηκε να στηθούν κυβερνήσεις μαριονέτες, το ίδιο και κυβέρνηση στη Δανία και δεν περιμένει κανένας τίποτα το ιδιαίτερο από την κυρία Τόρνινγκ Σμιτ αλλά η μόνη απέτηση που έχουμε εμείς είναι να έρχεστε τακτικά εδώ στις Βρυξέλλες, στο Στρασβούργο για να μπορέσουμε τουλάχιστον να αποφύγουμε την τεράστια καταστροφή που θα μπορούσε να προκληθεί στην Δανία. και φαίνεται ότι εσείς ενώ θα έπρεπε να παλέψετε για τη σωτηρία της Ευρώπης ε, παίζετε το, παίζετε το βιολί σας πάνω στο Τιτανικό ενώ βουλιάζει. Καλώς ήρθατε λοιπόν στην Ευρώπη κυρία μου με τους φίλους σας τον κύριο Βαν Ρομπόη, τον κύριο Μπαρόσο κανένας όμως δεν είχε όρεξη να σας δει εδώ. Πρόκειται για μία love story λοιπόν την οποία πρέπει να αντιμετωπίσουμε. Κύριε Μέστερ μπορείτε να βάλετε τα ακουστικά σας, σας παρακαλώ. Η κυρία Σίνκλερ θέλει να σας κάνει μία ερώτηση. Κυρία Σίνκλερ, παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Μία ερώτηση για τον συνάδελφο που είναι μέλος από τη Δανία για τον φόρο επί των χρηματοπιστωτικών συναλλαγών που ο Δανός Πρωθυπουργός, η Δανής Πρωθυπουργός είπε ότι θέλει να προκινήσει. Είπαμε ότι αυτό θα κοστίσει πολλές θέσεις εργασίας. Και ο προηγούμενος Πρωθυπουργός ε, χαρακτήρισε τον φόρο αυτό ανοησία. Τι έχετε να πείτε. Παρακαλώ κύριε Μέσσερ Σμιτ. Μα ένας ε, φόρος ε, επί των ε, συναλλαγών θα ήταν πάρα πολύ κακό πράγμα για, τον, για την ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης. Θα, θα επίση επίσης και την αγορά της εργασίας. και δεν ξέρουμε τελικά τι σκέφτονται οι Δανείοι για όλα αυτά θα έπρεπε να ρωτηθούν. Μάντλενερ για ένα λεπτό. Ευχαριστώ πρόεδρε. Δυστυχώς ε, κυρία Τόνινγκ Σμιτ ε, ποτέ δεν άκουσα τόσα άδεια ρητορική και τόσα κενά λόγια όπως αυτά που άκουσα από εσάς. Με το παρόσο μοιάζεται. Δεν λέει δεν λέτε τίποτα. Όπως έχουμε συνηθίσει από την Επιτροπή και από τον Παρόσο, εδώ και 15 χρόνια μας ε, υπόσχεται η Ευρώπη η οικονομική ανάπτυξη με τη συνθήκη της Λισαβόνας και όλα αυτά αποδείχθηκαν ανοησίες. Στην πραγματικότητα ο, Ευρωπαϊ... ο ευρωπαϊκός σοσιαλισμός οδήγησε σε μαζική ανεργία, σε οικονομική ύφεση και πολιτικές πρακτικές για να γεμίζουν οι λίγοι τις τσέπες τους. Να σας κάνω την εξή έκκληση στην Ολλανδία έχουμε ένα, μεγαλύτερα, ένα από τα μεγαλύτερα κοινωνικά συστήματα σε όλο τον κόσμο. Και είμαστε περήφανοι γι' αυτό, αλλά η ευρωπαϊκή γραφειοκρατία καταστρέφει αυτό το ολλανδικό σύστημα. Δεν είναι δυνατόν να έχουν οι ξένοι αλλοδαποί εργαζόμενοι να επωφελούνται μετά από ένα χρόνο δουλειά από το σύστημά μα. Θα πρέπει να διαρκεί τουλάχιστον 10 χρόνια αυτή η περίοδο. Είναι πάρα πολύ σημαντικό λοιπόν ε, η Ολλανδία να έχει τη δυνατότητα να αποκρούσει όλους τους Ρουμάνους και Βουλγάρους ε, τυχοδιώκτες για να διατηρηθεί το σύστημα της Ολλανδίας. Αν θα θέλατε λοιπόν, κυρία Χέλε Σμιτ, να το βάλετε αυτό στην κορυφή των προτεραιοτήτων σας. Ευχαριστώ. Τώρα το λόγο έχουν οι άλλοι ομιλητές. Μπέστε, για δύο λεπτά. Ε, ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα ήθελα να καλωσορίσω την ε, Δανική Προεδρία και ελπίζουμε ότι όλα θα εξελιχθούν για το καλύτερο και ότι θα υποστηριχθεί ευρύτατα. Ορισμένοι εκφράστηκαν κατά και όχι ικανοποιημένοι για την Δανέζικη Προεδρία η οποία όμως παρουσίασε εδώ τις προτεραιότητές της και έχουμε κατεπίγουσες υποθέσεις να αντιμετωπίσουμε στον τομέα της οικονομίας, το six pack και ελπίζουμε ότι η Δανία το επόμενο εξάμεινο θα σταθεί στο ύψος αυτών των προκλήσεων. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να, να έχουμε μια καλή προεδρία που θα μπορέσει να προχωρήσει στην ευρωπαϊκή ημερήσια διάταξη ξεπερνώντας τις διαφορές για την οικονομική κατάσταση η Δανία θέτει την προτεραιότητα στην ενεργειακή πολιτική. Πρόκειται για ένα ζήτημα πάρα πολύ σημαντικό και πρέπει να βρούμε μια γρήγορη λύση. Έχουμε 350 δισεκατομμύρια ευρώ τα οποία σπαταλούνται θα πρέπει να στον τομέα της ενέργειας θα πρέπει λοιπόν να προχωρήσουμε με μέτρα εξοικονόμησης στην ενέργεια. Οι Ευρωπαίοι εξαρτώνται κάθε μέρα και περισσότερο από τα πετρέλαια της Μέσης Ανατολής και το φυσικό αέριο του κυρίου Πούτινγκ. Μέσα από την οδηγία για την ενεργειακή αυτάρκεια θα πρέπει να παλέψουμε για την αυτάρκεια της Ευρώπης στον ενεργειακό τομέα, συμβάλλοντας στην οικονομική ανάπτυξη, στη δημιουργία θέσεων απασχόληση στον τομέα της ενέργειας. Η Δανία θα πρέπει να απαντήσει σε όλα αυτά τα ζητούμενα κατά το επόμενο εξάμεινο. Εγώ θα ήθελα η Δανέζικη Προεδρία να είναι θαραλέα, θαραλέα και στις στιγμές εκείνες που δεν έχουμε συνένεση για να προχωρήσουμε με σημαντικά αποτελέσματα. Ευχαριστώ. Δυόμιση λεπτά. Ο κύριος Γιώργενσεν. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ευχαριστώ την Πρωθυπουργό που μας παρουσίασε τις προτεραιότητες της Δανέζικης Προεδρίας για το επόμενο εξάμεινο. Εμείς θέλουμε να οικοδομήσουμε μια πιο ανταγωνιστική και πιο ασφαλή Ευρώπη ορίζοντας έναν αποφασιστικό δρόμο για την Ευρωπαϊκή Ένωση η Ευρωπαϊκή Ένωση θα μπορέσει να προχωρήσει πέρα από το πεδίο των συζητήσεων στο Στρασβούργο και στις Βρυξέλλες διότι η πραγματικότητα διαφέρει κατά πολύ στις χώρες μας. Ακόμη και αν οι αποφάσεις που λαμβάνουμε εδώ είναι αποφάσεις που έχουν τεράστιες επιπτώσεις για τους πολίτες μας, από την Κύπρο μέχρι το, την ε, Κοπεχάγη. Αλλά όταν μιλάμε εμείς για μια πιο δυναμική Ευρώπη, πρέπει να εννοήσουμε ότι θέλουμε να δημιουργήσουμε ανάπτυξη θέσης εργασίας και οι πολίτες μας μας ζητούν να προχωρήσουμε σε δίκαιες μεταρρυθμίσεις και αυτή η ισορροπία είναι δύσκολο να επιτευχθεί. Λίγο πολύ όπως ε, στις ιστορίες αγάπης που πρέπει κανείς να βρει την αδερφή ψυχή. Υπάρχουν περιπτώσεις όπως η Ελλάδα. Είναι πάρα πολύ δύσκολο να διαπραγματεύεται σήμερα κανείς με χώρες σαν την Ελλάδα. Το μήνυμα λοιπόν είναι ότι η Ευρώπη πρέπει να παραμείνει ενωμένη με ένα όραμα. Ένα όραμα που θα μας επιτρέψει να βγούμε από την κρίση. Εμείς ε, είμαστε στην πρωτοπορία για το κλίμα, για το περιβάλλον και σε αυτόν τον τομέα μπορούμε να δημιουργήσουμε ανάπτυξη για την ενεργειακή αυτάρκεια. Μπορούμε να προωθήσουμε ένα 2% επιπλέον. Αυτό θα δημιουργούσε 2 εκατομμύρια νέες θέσεις εργασίας. 2 εκατομμύρια Ευρωπαίοι άνεργοι θα μπορούσαν να βρούνε θέσεις εργασίας. Αλλά αυτό θα μπορέσουμε να το πετύχουμε μόνο αν είμαστε όλοι ενωμένοι. Καταπολέμηση της τρομοκρατίας, καταπολέμηση της εγκληματικότητας, διασυνοριακή εγκληματικότητα και σε αυτό θα πρέπει να είμαστε ενωμένοι συνεργαζόμενοι πέραν των συνόρων. Χρειαζόμαστε ένα πρόγραμμα με οράματα και φιλοδοξία. Καλή επιτυχία, Πρόεδρε. Δέχεστε σας παρακαλώ μία ερώτηση από τον κύριο Ντάρτμουν. Παρακαλώ. Κύριε Γιώργινσεν, έχετε συνειδητοποιήσει, έχετε σκεφτεί ότι οι πολιτικές της Κομισιόν δημιουργούν Ευρώπη τεράστιας ανεργίας. Εσεί έχετε σκεφτεί, αγαπητέ, ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν χαράζει πολιτικέ, ε, υποβάλλει προτάσει. Εσεί και εγώ δημορφώνω πολιτικέ. Και ο πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου είναι μέρο αυτή τη διαδικασία. Ε, και αν κάνουμε ακριβώ αυτά τα οποία η Ευρωπαϊκή, η Δανέζικη Προεδρία, συγγνώμη, έχει προτείνει, δηλαδή να στοχεύσουμε σε πολιτική ανάπτυξη η οποία να είναι αηφόρο και κοινωνικά φιλική, ούτω τότε θα κάνουμε τη διαφορά. Τότε θα έχουμε μια πολιτική ευμηνία για τους ε, Ευρωπαίους. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ρούντε για δύο λεπτά. Κυρία Πρωθυπουργέ, Καλώ ορίσατε εδώ που ξεκίνησατε τη διαδρομή σα και θα πρέπει να σα μιλήσω στα αγγλικά, διότι θα ήθελα να σα συγχαρώ εσά και την κυβέρνησή σα και τελευταία φορά το οποίο το έκανα αυτό. Είχαμε εδώ την Επίτροπο Ρέντινγκ. Όμω τη μετάφραση πέρασε ω επίκριση. Οπότε γι' αυτό σα τα λέω στα αγγλικά για να με καταλάβετε μια που αυτά τα οποία θα να πω επίση θέλω να τα ακούσουν και οι συνάδελφοι. Θέλω επίση να συγχαρώ την Δανέζικη κυβέρνηση για τρει λόγου. Πρώτα-πρώτα, μπράβο που αφού γκραστήκατε τη φωνή του Κοινοβουλίου όσον αφορά τι προτεραιότητε, τι κορυφές και για το ότι θα συνεχίσετε αυτό το οποίο ήδη βρίσκονται επί τη τραπέζη. Πρόκειται για κάποιο πρόγραμμα το οποίο είναι ε, φιλόδοξο, το οποίο όμω ταυτόχρονα είναι και ρεαλιστικό και αυτό αποδεικνύει ότι έχετε ξεκάθαρα καταλάβει το ρόλο σα και επίσης κατακλείδη εσεί και οι υπουργοί σα, κυρία Πρωθυπουργέ κάνατε, ε, τη, τη δουλειά σας, διαβάσατε το μάθημά σας και ήσασταν πάρα πολύ επιμελής ε, όσον αφορά ε, τη συνεργασία με το Κοινοβούλιο. Σας ευχαριστούμε και είμαι βέβαιος ότι η στήριξη την οποία επιζητείτε θα σας δοθεί. Όμως, όμως πριν... Πριν, πριν παρασυρθείτε κυρία Πρωθυπουργέ από όλα αυτά τα καλά μου λόγια θα ήθελα να σας απευθύνω και μερικές καυτές ερωτήσεις πρώτα-πρώτα ε, τι λέτε όσον αφορά αυτό το ναρκοπαίδιο το οποίο τώρα αναδύεται όσον αφορά τις διακυβερνητικές συμφωνίες και πώς θα αποφύγουμε τη διάσπαση της Ευρώπης. Δεύτερον, δεύτερον λέγω, τι πρεσβεύει η ιδανική κυβέρνηση για τον φόρο Τόιμπιν όσον αφορά τα τελευταία σχέδια της Κομισιόν. Είναι δυνατόν αυτό να μας ε, κοστίσει 130 ε, θέσεις απασχόλησης. Τελευταίο δε το εξής. Συζητούμε για την ε, επανένωση των ε, κανόνων που θα διεύουν την επανένωση των, οικογενειών και ε, ο κύριος Σούλτς απέσυρε αυτό το οποίο είχε διατυπωθεί με αυτό τον κανόνα των 24 ετών και εσείς λέτε ότι πρόκειται για ευκαιρία ή όχι και έτσι να ξεκινήσουμε τη δουλειά μας για να έχουμε ένα τέτοιο κανόνα και πάλι. Αυτές είναι οι ερωτήσεις μου. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας και καλή επιτυχία στο έργο σας. Δέχεστε μία ερώτηση από τον κύριο Κόνη. Μπορείτε να βάλετε τα ακουστικά σας παρακαλώ. Μπορείτε σας παρακαλώ να βάλετε τα ακουστικά σας. Δέχεστε μία ερώτηση από τον κύριο Κόνη. Συγγνώμη, συγγνώμη. Μία παρεξήγηση. Δεν ήθελε ερώτηση, απλώς ήθελε να μπει στον κατάλογο μιλητών για το Catch the Eye. Κυρία Τούρνεν, για ένα λεπτό. Καλώς ορίσατε, κυρία Πρωθυπουργέ. Σας ευχαριστούμε θερμά εκ μέρους της ομάδας μας Πρόκειται για έναν άνεμο, ένα νέο άνεμο το να βλέπει κανείς μια γυναίκα στην καθοδήγηση της Ευρώπης όπου βλέπουμε μόνο σκούρα ανδρικά κουστούμια. Είστε μία νότα δροσιάς. Είμαι ιδιαίτερα ικανοποιημένη που η Προεδρία έχει θέσει ως προτεραιότητα την υπέρβαση της ε, κρίσης. Εγώ πιστεύω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να δημιουργηθούν νέες θέσεις απασχόλησης για εκατομμύρια Ευρωπαίους που δεν έχουν σήμερα δουλειά, κυρίως τους νέους. Εμείς θα πρέπει να φανταστούμε <coughs> σήμερα ένα νέο συμβόλαιο μεταξύ των γενεών για να εγγυηθούμε ότι η ανεργία των νέων θα μειωθεί και οι νέοι Ευρωπαίοι θα μπορέσουν να βρουν μια δουλειά. Μόνο έτσι θα μπορέσουμε να βγούμε από την κρίση. Επίσης είναι θεμελιώδες να μπορέσουμε να είμαστε ενωμένοι για να υπερβούμε την κρίση. Δεν μπορούμε να συνεχίσουμε με αντιπαλότητες και καυγάδες μεταξύ ημών. Χρειαζόμαστε μια δίκαιη οικονομία εγώ σήμερα έτρεφα μεγάλες προσδοκίες για τη Δανέζικη Προεδρία και ελπίζω να επιβεβαιωθούν. Η κυρία Ρόσμπαχ για δύο λεπτά. Ευχαριστώ. Πρόεδρε, καλώς ορίσατε κυρία Πρωθυπουργέ. Η Δανέζικη Προεδρία πρέπει να αντιμετωπίσει αυτό το εξάμεινο τεράστιες προκλήσεις. Προσδοκούμε η Δανέζικη Προεδρία να επικεντρωθεί στην μεταρρύθμιση του τομέα της ενέργειας ε, στην Ευρώπη να ποντάρει στην ε, αυτάρκεια αναπτύσσοντας νέες πηγές ενέργειας ε, διότι η υδραυλική, η ηλιακή ενέργεια, η αιωλική ενέργεια δεν αρκούν πια. Η Δανέζικη Προεδρία έρχεται σε μία στιγμή ιδιαίτερα σοβαρή και κρίσιμη η ενέργεια πλήττει τους Ευρωπαίους, κυρίως τους νέους. Αυτή η τάση μπορεί να αλλάξει όμως αν στοχεύσουμε στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις οι οποίες αντιμετωπίζουν δύσκολες καταστάσεις. Πρέπει να ξαναξεκινήσει η ανάπτυξη. Δεν θα πρέπει η Προεδρία να συγκεντρωθεί στην τροποποίηση των συνθήκων πράγμα για το οποίο δεν ε, τρέφουν ιδιαίτερη συμπάθεια οι πολίτες χρειάζεται να λάβει μέτρα που θα έχουν συγκεκριμένα και αυτά αποτελέσματα χρειάζεται μεταρρύθμιση της γεωργικής πολιτικής χρειάζεται μεταρρύθμιση της, αλή, της πολιτικής αλίας σε μία φάση δημοσιονομικών περικοπών σε όλες τις χώρες ο ρόλος αυτού του Κοινοβουλίου είναι πάρα πολύ σημαντικός και για τη μεταρρύθμιση της ΚΑΠ και της πολιτικής αλίας. Αυτή η πολιτική είναι πανάκριβη σήμερα. Δεν μπορούμε εμείς ε, ε, να χορηγούμε αδιακρίτως επιδοτήσεις οι οποίες δεν έχουν κανένα θετικό αποτέλεσμα. Οι προτεραιότητες δυστυχώς της Δανέζικης Προεδρίας τους τους τομείς μας φαίνονται αφηρημένες. Ελπίζουμε να γίνουν πιο απτές κατά τους επόμενους μένους, μήνες. Ο Πολ Μάρφη για ένα λεπτό. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Τέσσερα χρόνια νιώθουμε στο πετσί μας την λιτότητα παντού στην Ευρώπη και τα αποτελέσματα είναι ξεκάθαρα. Έχουμε τώρα έναν αρνητικό κύκλο ε, οικονομικής εξέλιξης που έχει εφαρμοστεί και σε Ιρλανδία αλλά και σε Ελλάδα. Δεν μπορούν ε, ούτε, ούτε να δώσουν οι Έλληνες τα παιδάκια τους και τώρα ε, βρισκόμαστε μπροστά στο φάσμα της ε, ύφεση τώρα το 2012 και όμως όλοι μιλήσατε και ο κ. Μπαρόσο για ανάπτυξη όμως αν κανείς διαβάσει λεπτομερώς το πρόγραμμα το δεν συνιστά πολιτική ανάπτυξη αλλά λιτότητας Άρα θα πρέπει να δούμε τι θα γίνει με την οικονομική διακυβέρνηση. Πρόκειται για μία μέθοδο που παγιώνει αυτή τη λιτότητα παντού στην Ευρώπη. Ε, αυτό είναι, ο ορισμός της, της ε, παράνοιας, δηλαδή ότι κανείς να κάνει ο παρανοϊκός τι κάνει, κάνει το ίδιο πράγμα συνέχεια και περιμένει κάθε φορά να του προκύψουν διαφορετικά αποτελέσματα. Αυτό κάνετε και εσείς. Και αυτοί που ελέγχουν τα ομόλογα οικονομάνε στην πλάτη του και εμείς κάτι θα πρέπει να γίνει όσον αφορά αυτή τη συνθήκη της λιτότητας γιατί έτσι θα παγιωθεί αυτή η κατάσταση. Ε, μιλούμε τώρα για το δικαίωμα του Ιρλανδικού λαού για ελεύθερο δημοψήφισμα στο οποίο όμως να απουσιάζει η προεκλογική εκστρατεία που θέλει να επιβάλλει το ναι. Ευχαριστώ συνάδελφε. Για ένα λεπτό η κυρία Ζαμπέλα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κυρία Πρωθυπουργός, καλή επιτυχία το επόμενο εξάμηνο. θα ήθελα να κάνω δύο συγκεκριμένες προτάσεις ως προσθήκη ή βελτίωση στην ήδη υπάρχουσα πολιτική της επιτροπής. στον τομέα της ενέργειας θα μπορούσε η προεδρία σας να αναλάβει την πρωτοβουλία της καταγραφής όλων των υπαρχουσών πηγών ενέργειας στην ευρώπη. θα πρέπει να ξέρουμε τι πηγές ενέργειας διαθέτει η ευρωπαϊκή ένωση και ποιες δεν είναι ρεαλιστικές οι επενδύσεις που κάνουμε σε αυτήν. δηλαδή έχουμε φωτοβολταϊκά σε χώρες που δεν έχουν ήλιο καταγραφή των υπαρχουσών πηγών ενέργειας και δεύτερη πρωτοβουλία στον τομέα της απασχόλησης. η wall street journal yesterday είχε αφιέρωμα στη μεγάλη έξοδο του εργατικού δυναμικού από την ευρωπαϊκή ένωση. θα πρέπει να δούμε αυτή την αλλαγή στον ιστό της αγοράς εργασίας της ευρωπαϊκής ένωσης. είναι δύο πρωτοβουλίες στην ενέργεια και στην απασχόληση που σας προτείνω. ευχαριστώ. Ευχαριστώ κυρία Ευχαριστώ, Πρόεδρε, κυρία Πρωθυπουργέ. Ε, εύχομαι να αντιλαμβάνεστε ότι πολλοί κόσμος στην Ευρώπη έχει υψηλέ προσδοκίες από την Προεδρία σας, από την Δανική Προεδρία. Η χώρα σας ήταν από τα λίγα κρατημέλη που επέδειξε το θάρρος για να πάρει τα απαραίτητα προβλήματα για να περιορίσει το πρόβλημα της μετανάστευσης. Αυτό συχνά ε, το απαξίωσε και η Ευρωπαϊκή Ένωση και κάποιες κυβερνήσεις, αλλά το, η κυβέρνησή σας, το κράτος σας μάλλον, έλαβε θεραλές αποφάσεις και σε ό,τι αφορά το θέμα των ε, σκίτσων, σε ό,τι αφορά την Ισλαμική ε, έλλειψη ελαστικότητας. Ελπίζω και σε άλλα θέματα, κύριε Πρωθυπουργέ, να ε, υποστηρίξετε το δικαίωμα των χωρών να έχουν δική τους πολιτική για το άσυλο και τη μετανάστευση, γιατί σήμερα Υπάρχει κρίση στα εξωτερικά σύνορα του Σέγγεν, όπως και ευρω... ευρωπαϊκή κρίση. Ευχαριστώ συνάδελφε. Ο κύριος Λάγκεν για 1,5 λεπτό. Ευχαριστώ πρόεδρε. Θα ήθελα να συγχαρώ την ε, Πρωθυπουργό της Δανίας για το πρόγραμμά της είναι από δανεικής πλευράς κάτι εντελώς καινούριο για μας και θα κάνουμε τα πάντα για να υποστηρίξουμε ενεργά το πρόγραμμα αυτό και στην εφαρμογή των μεμονωμένων μέτρων, όπως για παράδειγμα στα δημοσιονομικά, αλλά και σε ό,τι αφορά τις προσπάθειές σας να μην περάσει η διακυβερνητική μέθοδος, αλλά η κοινωτική μέθοδος. Τονίσατε ότι θα τονίσετε αυτά τα στοιχεία. Σας υποστηρίζουμε αν προωθήσετε αυτές τις τις πρωτοβουλίες. Να προσθέσω το εξής. Ας βγει επιτέλους η Δανία με τη βοήθειά σας από τον ευρωσκεπτικισμό, από τη γωνία. Έχετε την ευκαιρία όχι μόνο να στραπήσετε το ευρώ, αλλά να αλλάξετε αυτή την δανεική κοινή γνώμη και να κάνετε ένα ενεργό βήμα προς το ευρώ. Και να προσθέσω και κάτι ακόμα. Το πρόγραμμά σας το υποστηρίζουμε, αλλά διάβασα σε πολλές περιπτώσεις ότι θέλετε να κάνετε ένα βήμα προς την Τουρκία. Σήμερα δεν αναφερθήκατε σε αυτό. Σας παρακαλώ, κυρία Πρωθυπουργέ. Κάντε μας τη χάρη κατά την εξάμεινη προεδρία σας και πείστε την Τουρκία προκειμένου να άρουν τους φραγμούς ε, για την Κύπρο, για την επόμενη Προεδρία. Αυτό θα είχε νόημα για την Τουρκία, γιατί αν θέλει να εξακολουθήσει να μπλοκάρει η Τουρκία την Κύπρο, σε τελική η ανάλυση μετά από έξι μήνες θα διαπιστώσετε ότι στο σημείο αυτό ενδεχομένως δεν επιτελέσατε όπως θα θέλατε τα καθήκοντά σας. Σας παρακαλώ φροντίστε το και θα σας υποστηρίξουμε. Ευχαριστώ κύριε Λάγκεν. Ο Κλοντ Μωράες για ένα λεπτό. Κυρία Πρωθυπουργέ, καλώς ορίσατε. Το Κοινοβούλιο. Με επιτρέψτε να σας πω πρώτα-πρώτα ότι σας καλωσορίζει, σας υποδέχεται η οικονομική κρίση και βέβαια ήμασταν δίπλα-δίπλα εδώ στην Κοινοβουλική Επιτροπή μας στο Κοινοβούλιο και ξέρω την αξία του έργου σας και ξέρω ότι ήσασταν ε, εδώ από νωρίς προετοιμασμένοι δεν διστάσατε μπροστά στις ε, προκλήσεις των διαφορετικών θεμάτων ε, ακόμα και για τα εσωτερικά και τη δικαιοσύνη ε, είναι κρίσιμη η καιρή και αυτό το οποίο εσείς επιτελέσατε είναι πολύ σημαντικό δεν διστάσατε, δεν δηλιάσατε και βοηθήσατε να έχουμε μια πάρα πολύ σωστή αρχή στην διαδρομή μας και οπότε θα πρέπει να δούμε τι θα γίνει με τα θέματα Schengen είναι κομβικό θέμα για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα τι θα κάνουμε με το άσυλο. Ε, <clears throat> τι θα για τα, ε, για, για, τα, για τα σχετικά και οπότε δεν μπορούμε να σας ευχαριστήσω και πάλι για το πόσο με θέσεις και συνεργάτε σας και για την Ουγγαρία επομένως να δούμε ε, μια στεναρή στάση από πλευρά τη Προεδρίας, γιατί εκεί διακυβεύονται κάποια θέματα κοινοτικών αξιών. Βέβαια έχουμε και την χρηματοπιστωτική κρίση που και αυτό είναι στο επίκεντρο των προσπαθειών μας. Ευχαριστώ κύριος Λάμστορφ. Κυρία Πρωθυπουργέ, να ξεκινήσω λέγοντας ε, ότι σας ευχαριστώ. Μα μπλε κάρτα. Υπάρχει έτοιμα και μπλε κάρτα. Ε, Κύριε Μωράες. Ε, Αν συμφωνεί ο κύριος Μωράες θα κάνουμε μία εξαίρεση. Παρακαλώ. Σας ευχαριστώ. Κύριε Μωράες, είπατε ότι επιθυμείται η Δανέζικη Προεδρία να αντιμετωπίσει τα θέματα που ανέκυψαν στην Ουγγαρία. Γι' αυτό το κάνει κατεπηγόντως και αποφασιστικά. Το εμείς, τι πάνε να πει κύριε Μωράς, ποιο ποσοστό των ψηφοφόρων σας θεωρείτε θα επιθυμούσαν η Προεδρία να ασχοληθεί με την Ουγγαρία τώρα, ενώ σοβεί αυτή η τρομερή κρίση στην Ευρώπη και έχουμε ανεργία, αυτό. Πόσοι, πόσοι πόσοι από τους ψηφοφόρες σας, τι ποσοστό είναι αυτό το οποίο απαιτεί το να ασχοληθούμε με το συνταξιοδοτικό όριο στην Ουγγαρία και γενικά τα, τα επιμέρους ε, μέτρα της ε, Ουγγρικής κυβέρνησης. Μωράς, ακούστε τι είπα. Είπα ότι είναι κομβικό θέμα για μας και για την Προεδρία η χρηματοπιστωτική κρίση. Προσέξτε. Βεβαίω και δικαιούμαι από το καταστατικό να υποβάλλω το θέμα για την Ουγγαρία. Είναι το διακύβευμα η αξία της Ένωσης. Ναι, μας προβληματίζουν αυτά τα θέματα. Και αυτό που ανέβησαν στην Ουγγαρία δεν είναι θέματα που αφορούν μόνο τον Ουγγρικό λαό. Είναι η πολιτική της κυβέρνησης και οποιαδήποτε κυβέρνηση που θίγει βασικές ε, αξίες, τότε αυτό μας απασχολεί, πρέπει να μας απασχολεί όλου. Φυσικά και δεν είναι το μόνο θέμα το οποίο είναι σημαντικό και το οποίο απαιτείται να συζητηθεί στο Κοινοβούλιο. Πρόεδρο. Δύο λεπτά κύριε Αλεξάνδρ Λάνστορ. Ευχαριστώ πρόεδρε δεύτερη απόπειρα. Ξαναξεκινάω. Θα ήθελα καταρχά να σα ευχαριστήσω μετά την ανάληψη των ε, πρωθυπουργικών σα καθηκόντων. Ε, καταργήσατε τι προηγούμενε ιδέες, τι προηγούμενε. Ε, ε, ιδέε τη κυβέρνηση, τη προηγούμενη κυβέρνηση, για να ξαναμπούν σύνορα μεταξύ Ιρμανίας και Δανία, μεταξύ Σουηδία και Δανία. Ήταν πολύ καλή η είδηση αυτή για τι επιχειρήσει, για του πολίτε, για τι μεταφορικέ εταιρείε ιδιαίτερα και των δύο χωρών. Σα ευχαριστώ πάρα πολύ. Ήταν πάρα πολύ καλά τα μέτρα αυτά. Δεύτερο σημείο και θα συμφωνήσω με τον Βέρεν Λάγκε. Είναι σας παρακαλώ να προσπιστείτε την κινητική μέθοδο. Νομίζω ότι σε διάφορες περιπτώσεις ζήσατε το τι σημαίνει να ξανακυλήσουμε στον ε, διακυβερνητισμό του 19ου αιώνα και στην όλη νοοτροπία αυτά που υποστηρίζει ο κύριος Σαρκοζή. Αν αυτός είναι ο νέος τόνος, θα πρέπει να αναγνωρίσουμε ένα επιπλέον επιχείρημα υπέρ του, της διακοινωτικής μεθόδου. Είπατε ότι θα πρέπει να υπάρχει μια ενιαία εικόνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς τα έξω καλό θα είναι να αξιοποιήσουμε την ευκαιρία της Προεδρίας σας για να ξεκινήσει μια συζήτηση για το κατά πόσο θέλουμε να διατηρήσουμε την πολιτική άμυνας και ασφάλειας. Όλοι συμμετέχουν στην πολιτική αυτή, εκτός από την Δανία. Τελευταίο σημείο. Η ομάδα μου μαζί με τους πράσινους και τους σοσιαλδημοκράτες θέλουμε να ξεκινήσει τη διαδικασία βάση του άρθρου 7 παραγράφου 1 κατά της Ουγγαρίας, αλλά το Συμβούλιο είναι αυτό που θα πρέπει να λάβει τα μέτρα αυτά. Σας ε, καλώ να οργανωθείτε, να συγκεντρωθεί η πλειοψηφία των 4 πέμπτων στο Συμβούλιο για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε το θέμα της Ουγγαρίας. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ αγαπητέ συνάδελφοι. Ο κύριος Τούρμες για ένα λεπτό. Αγαπητή ε, κυρία Πρωθυπουργέ, αποτελέσματα. Αυτό θέλουμε. Δεν αμφισβητούμε τις προθέσεις σας και είμαι ο εισηγητής του ψηφίσματο μας, του κειμένου μας για την αποτελεσματική χρήση ενέργειας και οπότε αυτό με απασχολεί όμως σήμερα θέλω να θίξουμε κάτι το οποίο νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό και γι' αυτό και θα πρέπει ε, βράχει πρόθεσμα να ελκύσουμε κάποιε επενδύσει. Δηλαδή, πρόκειται για την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, η οποία το Δεκέμβριο του 2008 ε, απεφάσισαν σχετικά με εκείνη 27 κυβερνήσεων ότι το 2009 θα αυξήσουν το κεφαλαιό από 55 σε 80 δις. Το 2009 το απεφάσισαν αυτό. Προσέθεσαν δηλαδή οι 25 δις τα οποία θα επενδύονται σε συγκεκριμένα προγράμματα και σε κάποιο είδου εταιρικά ομόλογα τα οποία θα διάσωζαν, θα προστάτευαν τέλο πάντων τη βιομηχανία σήμερα. Έχουμε την πιστοτική κρίση. Και η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων για του χρόνου έχει μειώσει τι επενδύσει τη. Τι κατέβασε στα 60 δι. Επομένω, τι γίνεται, γιατί με την σημερινή συγκυρία κάνουμε αυτό το πίσω γύρισμα και κόπηκαν αυτά τα 20 δι όσον αφορά δηλαδή τις επενδύσεις που θα κάνει και την επενδυτική δυνατότητα και για πες μας γιατί η ΕΤΕ δεν αξιοποιεί αυτό το, το, το, το, οποίο είπε για τις ιδιωτικές τράπεζες ο κύριος Δράγκη. 500 δις είπε ο κύριος Δράγκη. Έχουν οι ιδιωτικές τράπεζες τα οποία όμως τα πάνε στην ιδιωτική τράπεζα. Δεν τα πάνε ε, τα, χρήματά τους στην πραγματική οικονομία. Ε, πρόκειται για το 1%. Αυτά τα 80 δις, τα οποία το 2012 θα πρέπει να πάνε σε ευρωπαϊκή οικονομία. Νομίζω ότι αυτό θα τόνωνε πάρα πολύ την οικονομία και αυτό το αυτό έκανε κιόλας και κεραυνοβόλα. Ευχαριστώ. Η Μάρα Μπιτσότο έχει το λόγο. Η Ευρώπη γκρεμίζεται Και η Δανέζικη Προεδρία υπόσχεται απόλυτη εμπιστοσύνη στην ευρωπαϊκή μοίρα και θέλει να δράσει ως τσομπανόσκυλο της ευρωγραφειοκρατίας και του Συμβουλίου. Δεν συμφωνώ με αυτά. Εγώ δεν καταλαβαίνω πώς μπορούμε σήμερα να θεωρούμε προτεραιότητα την διεύρυνση σε βαλκανικές χώρες. Μα υπάρχουν άλλα προβλήματα να αντιμετωπίσουμε για το πώς θα ενσωματώσουμε, από το πώς θα ενσωματώσουμε νέες χώρες. Τουρκία. Η Δανία εξωθεί για την προσχώρηση της Τουρκίας. Ευτυχώς που η Τουρκία δεν προσεγγίζει τις παράμετρους για να γίνει μέλος, αλλά το παράδοξο ποιο είναι, Στη φάση που το ευρώ βρίσκεται σε ρίσκιο πτώχευσης, η Δανέζικη Προεδρία θα πρέπει να τη σώσει. Βέβαια, η Δανία βρίσκεται εκτός ευρώ, γιατί για το, από το ευρώ δεν είχε ποτέ εμπιστοσύνη. Ευχαριστώ και τώρα η κυρία Σινκλέρ. Για ένα λεπτό έχει το λόγο. Κυρία Πρωθυπουργέ, ξεκινάτε την Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης όπου ε, υπάρχουν απαράτακτες ε, νοτροπίες στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είδαμε πρόσφατα ότι ελεγμένοι ηγέτες ε, εκδιώχθηκαν και αντικαταστάθηκαν από τεχνοκράτες που δεν έχουν εκλεχθεί. Με μια ενδεχόμενη νέα συνθήκη, ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός προσπαθεί να συνενώσει υπό αμφίβολες δημοκρατικές συνθήκες τα 27 κρατημέλη. Και η Ευρωπαϊκή Ένωση στρέφει το βλέμμα της. Αναλαμβάνετε λοιπόν τα καθήκοντά σας σε μια κρίσιμη στιγμή, σε μια στιγμή ενδεχόμενης ε, εξαφάνισης του, ευρώ. του ευρώ. Χρειαζόμαστε ισχυρή ηγεσία. Πώς είναι δυνατόν όμως ε, να το αναλάβει αυτό μια χώρα εκτός του ευρώ και η Ευρωπαϊκή Ένωση στρέφεται προς το Διεθνές ε, Νομισματικό Ταμείο. Το Ηνωμένο Βασίλειο που είναι εκτός Ευρωπαϊκού του ευρώ να συμμετάσχει. Ευχαριστώ. Ο κύριος Μάουρο για 1,5 λεπτό έχει το λόγο. Μάριο Μάουρο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κυρία Πρωθυπουργέ, στο πρόγραμμα που μας αναφέρατε διαφαίνεται ότι η πρώτη προτεραιότητα της Δανέζικης Προεδρίας είναι να εγγυθεί μια υπεύθυνη ευρωπαϊκή οικονομία. Τι σημαίνει αυτό? Μια Ευρώπη πιο υπεύθυνη που θα έχει μεγαλύτερη συνέστηση του κινδύνου που την περιμένει. Το μεγαλύτερο εμπόδιο σήμερα όμως είναι η ευρωπαϊκή leadership, η ευρωπαϊκή αρχηγία, όχι το ευρώ. Διότι είναι χώρες οι οποίες δεν ναι μεν συμμερίζονται το νόμισμα, αλλά όχι την leadership η ακινησία, η απραξία είναι το πρόβλημα των αρχηγών μας που πλήττει κυρίως τις χώρες που χρειάζονται αυτή τη βοήθεια. Χαιρετίζω κατά συνέπεια και την προσπάθεια της Πολωνικής Προεδρίας η οποία δεν ξέχασε ποτέ ότι βασικός στόχος είναι η ενότητα. Το μόνο όπλο που μπορεί να εξορκίσει το κακό. Διότι όλα τα υπόλοιπα αν δεν υπάρχει ενότητα είναι κάτι το οποίο μας ρίχνει στα μάτια του υπόλοιπου κόσμου και των πολιτών μας. Θέλω κύριε Πρόεδρε Σούλτς να σας συγχαρώ για την εκλογή σας και να σας πω ότι σημερίζομαι απόλυτα αυτήν την κοινοβουλευτική διάσταση που θέλετε να δώσετε στην Ευρώπη. Η κυρία Στρέλα για δύο λεπτά. Presidente, seja bem-vinda, Senhora Primeira-Ministra, à União Europeia dividida entre os Estados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 της ομιλίας του κυρίου Μπαρόσο και της κυρίας Πρωθυπουργού, αλλά θα ήθελα να αντισταθώ σε αυτή την αγανάκτηση που επικρατεί σε ό,τι αφορά την ε, Ουγγαρία και σε ό,τι αφορά την ε, αντίδραση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Μου θυμίζει εμένα ως Αυστριακό το 2000 με τα ανόητα μέτρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά της Αυστρίας. Αμάυρωσε την εικόνα της. Αυτή η κίνηση είναι λανθασμένη. Η κυβέρνηση Ορμπάν ε, έχει αποδείξει επανειλημμένα ότι είναι δημοκρατική. Έχει εκλεχθεί από τα δύο τρίτα του γκρικού λαού. Το Συμβούλιο θα πρέπει να είναι αξιόπιστος ε, εταίρος και στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στο ΝΑΤΟ. Η Ουγγαρία δεν μπορεί να τη χάνει τέτοιας μεταχείρισης και όλοι όσοι οι φιλελεύθεροι, οι σοσιαλιστές που αγανακτούν Ευχαριστώ, διακόπτη ο Πρόεδρο. Και τώρα το λόγο έχει ο κύριος Όντι για 1,5 λεπτό. Σχετικά με τα οικονομικά και δημοσιονομικά, κύριε Πρωθυπουργέ, είπατε ότι η Δανία δεν θα ε, ε, δεν θα εμποδίσει την ολοκλήρωση στην Ευρωζώμη Τι σκοπεύετε να κάνετε όμως με τη μεταρρύθμιση του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης. Χρειαζόμαστε αυτό το κείμενο. Εμεί έχουμε και νέες πολιτικές πλειοψηφίες για, τον φόρο, για την επιβολή του φόρου στις, στη διακινήση του κεφαλαίου. Τώρα, η Κομισιόν θα πρέπει να διαπραγματευτεί εκπροσωπώντας ε, την Ένωση και εμείς ως Κοινοβούλιο θα πρέπει να συμμετέχουμε στη διαπραγμάτευση των εμπορικών συμφωνιών. Πρέπει όμως εμείς να είμαστε ιδιαίτερα ευφύεις να μην να, να, μην αφήσουμε να μας εξαπατήσουν. Πρέπει να προσέξουμε ιδιαίτερα τις συμφωνίες με τη Μερκοσούρ. Εσείς είστε μέλος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Ο πρόεδρος Σούλτς θέλει να προσκαλείτε στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Θα μας υποστηρίξετε ως προς την παρουσία του Προέδρου μας στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και την και, και, και ένα συμβούλιο το οποίο είναι αφιερωμένο μόνο στην ανάπτυξη. Καταλήν Ιβαν για ένα λεπτό. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Κυρία Πρωθυπουργέ, όλες οι φιλοδοξίες σας και οι στόχοι σας είναι ευπρόσδεκτοι, αλλά δεν πρόκειται να έχουν σημασία εκτός κι αν καταδικάσουμε τις τρέχουσες πρακτικές στην Ουγγαρία και στη Ρουμανία. Θα πρέπει να προσέξουμε να μην βλάψουμε ε, επιπλέον τον κόσμο του οποίου τα δικαιώματα πλήττονται. Θεωρώ ότι θα πρέπει να συζητήσουμε το τι συμβαίνει στη Ρουμανία, τι συμβαίνουν στην Ουγγαρία. Νομίζω ότι η Ευρώπη έχει λόγο ύπαρξη μόνο εφόσον πρόσπιζεται τη δημοκρατία και θα πρέπει να υπάρχει δημοκρατία και στα 27 κράτη-μέλη. Ευχαριστώ. Ο κύριο Ζάλμπα Πιτέγιν Νταΐν. 1,5 λεπτό. Κύριε Ζάλμπα. Ευχαριστώ και συγχαρητήρια κύριε Πρόεδρε. Κυρία Πρωθυπουργέ, εμείς ε, συζητάμε τις αποφάσεις του προηγούμενου Συμβουλίου και ελπίζουμε να μην μείνουν λόγια όλα αυτά και να υλοποιηθούν το συντομότερο. Είναι απαραίτητο να στείλουμε ένα μήνυμα προς τις αγορές, ένα αξιόπιστο μήνυμα. Μέχρι τώρα οι αγορές δέχονται ευνοϊκά τα μέτρα. Και θα πρέπει να συνεχίσουμε με την συνεργασία και την καλή θέληση που έχουμε δείξει μέχρι τώρα για τους επόμενους μήνες. Θα πρέπει σίγουρα να υπάρξει λιτότητα η οποία όμως θα συνοδεύεται από άλλα μέτρα που θα δημιουργούν ανάπτυξη και απασχόληση. Μόνο με τη λιτότητα δεν πρόκειται να βγούμε από την κρίση. Θα πρέπει να προχωρήσουμε σε μεταρρυθμίσεις, όχι μόνο σε συζητήσεις η Ισπανία έχει δεσμευτεί απόλυτα με αυτή την ιδέα. Γι' αυτό λοιπόν υποστηρίζουμε τις διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις που θα πρέπει να ληφθούν από τα κράτη-μέλη. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα από τη μεριά της παίρνεται θαραλέα όταν πρέπει να λάβει αποφάσεις. Πρέπει όμως να συμμετέχει και πιο δυναμικά στις δευτερογενείς αγορές του χρέους. Επίσης θα πρέπει να στήσουμε μηχαν, κοινούς δημοσιονομικούς μηχανισμούς. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Κύριε κυρία για ένα λεπτό. Ευχαριστώ. Κυρία Πρωθυπουργέ. Ευχαριστώ Πρωθυπουργέ. Σύμφωνα με τις ε, έρευνας, ε, η Δανία είναι το μικρόφωνο της ομιλητρίας είναι κλειστό. Μάλιστα. Μου πείτε το, το μικρόφωνο ο συνάδελφος από τη Δανία. Σύμφωνα με τις έρευνες λοιπόν, η Δανία έχει το μεγαλύτερο ποσοστό χαρούμενων, ευτυχισμένων ανθρώπων και θα ήταν καλό στην Προεδρία σας να... Φροντίσετε να βελτιωθεί η κατάσταση σε μια Ευρώπη δυστυχία. Συνήθω η Προεδρία έχει τόσες πολλές προτεραιότητες που στην τελική ανάλυση δεν υπάρχει καμία προτεραιότητα. Και το ίδιο συμβαίνει και με όλα τα θέματα τα οποία υπάρχουν στην Ευρώπη και τελικά υπάρχει τάση να ξεχνούνται. Τώρα μιλάμε για τον, την ενεργό γύρανση και αυτό αποτελεί βασικό ζήτημα και από οικονομικής άποψης. Θα πρέπει να διασφαλίσουμε ότι θα υπάρχει δυνατότητα σταδιοδρομίας για κάθε άτομο. Αυτό έχει να κάνει και με την ανθρώπινη αξιοπρέπεια αλλά και με την οικονομία. Είναι γεγονός ότι η ηλικία και η, η διακριτική μεταχείριση βάση της ηλικία είναι μια τάση που επικρατεί. Ενώ υπάρχουν εξαιρετικά παραδείγματα. Helmut Schmidt, Delors, ε, άτομα που ε, ε, λειτουργούν. Και πρόεδρο, η κυρία Γκάλ Πέλτ, για 1,5 λεπτό. Κυρία Πρόεδρε, παίρνετε σκητάλη σε αυτή την πάρα πολύ κρίσιμη συγκυρία. Όμω μπορείτε να αντιμετωπίσετε αυτέ τι δυσκολίε και έτσι δεν μπορεί να μπορέσετε να χειριστείτε αυτή την πρόταση η οποία προέρχεται από του συναδέλφου σοσιαλιστέ. Και γι' αυτό θα πρέπει να προσέξετε όσον αφορά το να μπει στο στόχο η Ουγγαρία. Εγώ δεν νομίζω ότι θα πετύχουν αυτά τα εγχειρήματα, διότι πριν από ένα χρόνο η Ουγγρική Προεδρία είχε καθορίσει έναν στόχο. Δηλαδή, είχε πει ότι θα πρέπει να γίνει συντονισμό των ευρωπαϊκών πολιτικών όσον αφορά κυρίω την οικονομική πολιτική και θα πρέπει να γίνει συντονισμό σε κλίμακα πανευρωπαϊκή. Εσεί. μπορείτε να συνεχίσετε ε, αυτή τη διαδρομή. Είμαι Ουγγαρέζα και ξέρω τι πάει να πει το να δουλεύει κανένας με βάση κοινέ ευρωπαϊκές πολιτικές και γι' αυτό και θέλω να συνεχιστεί η οικονομική διακυβέρνηση για να παρακολουθήσετε την πολιτική αυτή από κοντά οπότε θα πρέπει με, με, με διάβγεια να ασχοληθείτε με το θέμα αυτό επίσης δεν μπορούμε παρά να σας ευχαριστήσουμε για το ότι θα πρέπει να προσέξετε για τον άνθρωπο, όχι μόνο τα νούμερα όσον αφορά την οικονομική πολιτική. Δεν θα πρέπει να βάζουμε τα κράτη-μέλη σε δύο διαφορετικές κατηγορίες, τους καλούς και τους κακούς μαθητές. Όλοι, όλα τα κράτη-μέλη προσπαθούν. Οπότε σας εύχομαι καλή δουλειά, συνεχίστε με επιμονή στο έργο σας. Κύριε ένα λεπτό. Χαίρομαι κύριε Σούλτς που είσαστε ε, πρόεδρος γιατί έχουμε και πρωθυπουργό και πρόεδρο Σοσιαλδημοκράτε, σα ευχαριστώ. Λοιπόν, χαίρομαι πολύ που είστε εδώ πέρα, κυρία Σμιτ. Και ας πιστέψουμε στο θαύμα αυτό το επερχόμενο. Γιατί είναι τόσο δύσκολο το έργο, γιατί θα πρέπει να διατηρήσουμε την ένωση της Ευρώπης και η κρίση του ευρώ μας διχάζει. Θα πρέπει να πολεμήσουμε τους ευρωσκεπτικιστές, τους εξτρεμιστές δεν χαίρονται πάρα πολύ για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα πρέπει να, εφαρμόζουμε, να εφαρμόσουμε το πακέτο των έξι οδηγιών, να πάρουμε δύσκολε αποφάσει και υπάρχουν συμφαντικέ αμφιβολίε και σε μια χώρα που γνωρίζω καλά. Ωστόσο, υπάρχει ένα συνοπτικό πρόγραμμα της Προεδρία για μια δυναμική και ασφαλή Ευρώπη τονίζεται τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Χαίρομαι λοιπόν και είμαι βέβαιη ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα συνεχίσει το έργο της προκειμένου να γίνονται σεβαστές οι αξίες μας παντού. Και επιτέλους έχουμε μια ε, κυβέρνηση της οποίας ηγείται μια γυναίκα. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ και κόβει ο πρόεδρος του μικρόφωνο της Αμεριτρίας. Ευχαριστώ πολύ και τώρα ο κύριος Κάρας για 1,5 λεπτό και συγχαρητήρια για την εκλογή σας ως αντιπρόεδρος. Ευχαριστώ πρόεδρε και εσάς σας συγχαίρω. Χαίρομαι και προσβλέπω σε μια καλή συνεργασία. Η Προεδρία του Συμβουλίου έχει δύο προτεραιότητες. Ως στόχο έχει λοιπόν να ηγηθεί μιας Ευρώπης υπεύθυνη, Μιας Ευρώπης υπεύθυνη, δηλαδή μιας Ευρώπης δημοκρατικής. Τι προϋποθέτει αυτό, ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα πρέπει να συμμετάσχει σε κάθε απόφαση σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Χωρίς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν θα πρέπει να, γίνει καμία, να ληφθεί καμία απόφαση επί δανεικής προεδρίας. Κατά δεύτερον, μια υπεύθυνη Ευρώπη θα πρέπει να ενώνει, όχι να διχάζει. Ίσως είναι καλό το ότι δεν είσαστε στην Ευρωζώνη, γιατί γίνονται απόπειρες σήμερα να προκληθούν περαιτέρω διχασμοί. Όλα τα μέτρα που δίδονται ως απάντηση στην κρίση θα πρέπει να είναι κοινά μέτρα και θα πρέπει να οδηγήσουν στην ενοποίηση, στην πολιτική, την οικονομική και την δημοσιονομική. Και το δεύτερο σημείο προτεραιότητας θα είναι η ρύθμιση των χρηματοπιστωτικών αγορών. Σας παρακαλώ, μαζί με εμά στο Κοινοβούλιο, να προσπαθήσετε αμελητή να παρεμποδίσετε τα μεμονωμένα συμφέροντα και να ενισχύσουμε τα κοινό συμφέρον για την ρευστότητα, για την ε, διατήρηση του οικονομικού οικοδομήματος στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχουμε πάρα πολλά να κάνουμε. Μόνο μαζί θα τα πετύχουμε. Συγχαρητήρια κύριε Πρωθυπουργέ. Μπράβο σας για το πρόγραμμά σας. Έχει βέβαια κάποιο πασπάλιμο σοσιαλδημοκρατίας. Καταλαβαίνουμε πάντως τι θέλετε να κάνετε και θα πρέπει να προσέξουμε να μην έχουμε τον διχασμό που κινδυνεύουμε να έχουμε στην Ευρώπη σε σχέση με αυτό το οποίο θα πετύχουμε, δηλαδή την οικονομική σταθερότητα. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να το πετύχουμε και είναι πάρα πολύ σημαντικό το ότι η Προεδρία θα πρέπει να καταφέρει να κάνει ό,τι, ό,τι, ό,τι περνάει από το χέρι του, ώστε ενωμένη η Ευρώπη να προχωρήσει έτσι, ενωμένη. Να ξεκινήσει ένα κύμα μεταρρυθμίσεων για την εσωτερική ελεύθερη αγορά. Αλλά όλα αυτά, επαναλαμβάνω, με την Ευρώπη ενωμένη τόσο ώστε να ανακάμψουμε, να ξαναβρούμε το δυναμισμό μα. Αυτό θα είναι πάρα πολύ βασικό, θα είναι στο πήγαινο τη Δερμηνία και και γι' αυτό σα ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και ευχαριστώ και για να κλείσει η ομιλία αυτή, η συνάδελφο Κάριντ έχει το λόγο για ένα λεπτό. Αξιότιμοι συνάδελφοι, η επόμενη Προεδρία αντιμετωπίζει όντω μεγάλε προκλήσει στην κρίση του ευρώ, το πολιτέ δημοσιονομικό πλαίσιο, αλλά παράλληλα θα πρέπει να δώσουμε την απαραίτητη προσοχή στον ενεργειακό τομέα, ο οποίο καθίσταται όλο και πιο σημαντικό από γεωπολιτική άποψη και ειδικότερα θα πρέπει να προωθήσουμε την κοινή ενεργειακή πολιτική της Ένωσης. Θα πρέπει να προωθηθεί. Έχουμε νόμους οι οποίοι ορίζουν ότι το σύστημα διανομής διαχωρίζεται από την παραγωγή και εκ παραλλήλου υπάρχουν κρατημέλη που συνάπτουν συμβάσεις με τρίτες χώρες για αποκλειστικές τιμές για την παροχή ενέργειας εκτός της σχετικής νομοθεσίας της Ένωσης. Θα καλούσα λοιπόν την ε, Προεδρία της Δανίας να εξασφαλίσει ότι οι φυστάμενοι νόμοι δεν εφαρμόζονται μόνο στο εσωτερικό της Ένωσης, αλλά και στο εξωτερικό. Ευχαριστώ, λέει ο Πρόεδρος, Catch the Eye. Πάμε στη διαδικασία Catch the Eye. 28 άτομα σύγχυσαν το λόγο, προφανώς όμως δεν θα μπορέσω να τους δώσω σε όλους το λόγο έχουμε περίπου πέντε δυνατότητες, δυνατότητα για πέντε άτομα να λάβουν το λόγο. Θα προσπαθήσω να υπάρχει ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών και μεταξύ ομάδων. Ο κύριος Καργάνη έχει το λόγο πρώτος. Κύριε Πρόεδρε, εγώ πρέπει να πω ότι χθες και σήμερα ακούσαμε τρεις λόγους οι οποίοι είναι θερέλπιδες για την Ευρώπη. Τρία προγράμματα και τρεις στρατηγικές. Θέλω να πω στην Πρωθυπουργό ότι τα δύο πράγματα τα οποία είπε πολύ σημαντικά. Ότι η Δανία ακολουθεί τη μοίρα της Ευρώπης. Αυτή δεν είναι μια φράση στον αέρα. Είναι μια φράση που τη δεσμεύει να δυναμώσει την Ευρώπη, να κάνει ό,τι μπορεί για να υπερισχύσει η κοινοτική μέθοδος. Εμείς αντιμετωπίζουμε μια πολύ δύσκολη κατάσταση και δεν είναι ρητορική ερώτηση. Έχει διακοπεί η διαδικασία ανάπτυξης, της κοινοτικής ανάπτυξης. Και δεν έχουμε τροποποίηση των συνθήκων, αλλά συμφωνία μεταξύ των κρατών πρόκειται εδώ για διακυβερνητική διαδικασία η οποία εμποδίζει την ανάπτυξη και την εξέλιξη. Ευχαριστώ Παρακαλώ, κύριε Καρκάνη. Επόμενος ομιλητής η κυρία Κομές. Την προηγούμενη Παρασκευή και 13 οι ε, ευρωπαϊκοί ηγέτες αναφέρθηκε στα μέσα ενημέρωσης ότι είναι ανίκανοι να αντιμετωπίσουν την κρίση. Οι σοσιαλδημοκράτες υποστηρίζουν ότι τα προβλήματα προέρχονται από την ανταγωνιστικότητα μεταξύ της περιφέρειας και του πυρήνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα οίκια αξιολόγηση δεν συμφώνησαν με την προοδευτική αριστερά, αλλά η λιτότητα που υποστηρίζει η κυβέρνηση Μέρκελ και άλλες κυβερνήσεις ε, το μόνο που έχει ως αποτέλεσμα είναι ύφεση και επανάσταση στους λαούς της Ευρώπης. Ο φόρος από το συναλλαγό αποτελεί μια καλή αρχή, αλλά δεν αρκεί. Κοιτάξτε την Πορτογαλία. 19 από τις 20 σχετικές εταιρείε έχουν φύγει και έχουν μεταφέρει την έδρα τους ε, όχι για να διακόψουν, όχι για να ε, εξέλθουν του προλογικού καθεστώτος τους. Ευχαριστώ, λέει ο Πρόεδρος, η κυρία Λάτφορντ. Um, Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Πρώτα-πρώτα, ε, χαιρετίζουμε την προτεραιότητα που προσδίδει η Προεδρία στις χρόνιες ασθένειες και συγκεκριμένα ή στον διαβήτη. Και ε, ο συμπρόεδρος της Επιτροπής μας επίσης έχει ε, δηλώσει ότι θα δεσμευτεί να ασχοληθεί με τον διαβήτη που έχει σταματήσει νερολογική βόμβα, ότι έχει εξωτερωθεί, γιατί είναι τεράστιο το, το, κόστος για την κοινωνία αυτής της ε, ασθένεια. Παρακαλούμε την, την Δανέσκη Προεδρία να ασχοληθεί με μια πανευρωπαϊκή στατική κατά του διαβήτη. Επίσης θέλουμε να δούμε κατά πόσον η κυρία Πρωθυπουργός θα απαντήσει στην ερώτηση του Γκίφερ Χόφστατ. Τι κάνει το Συμβούλιο ούτω ώστε να εγκαλέσει την ε, Ουγγαρία να πάρει πίσω αυτές τις ε, απειλές που έχουν αναδειχθεί εκεί κατά των ευρωπαϊκών αξιών, κατά της δημοκρατίας. Ε, τι θα γίνει με, με, με την παραδοσιακή διπλωματία του Συμβουλίου που κανείς από τους κεφτά δεν κάνει τίποτα, κανείς δεν μετακινείται, διακόπτει ο Πρόεδρος. Παρακαλούμε, κάντε κάτι και αλλάξτε αυτή την ε, παθητική πολιτική παράδοση του, του, του, του Συμβουλίου. Επόμενο κυρία Πρωθυπουργέ, η Δανία τώρα με τη σειρά της αναλαμβάνει την ε, Προεδρία. Είπε ότι θα προσπαθήσει να βρει διέξοδο σε αυτή την κρίση. Μέσα σε ένα εξάμεινο. Σας πενθυμίζω επίσης ότι και η Βελγική και η Πολωνική Προεδρία είχαν τάξει παρόμοιες προτεραιότητες. Όλοι οι Ευρωπαίοι ενδιαφέρονται, αγωνιούν ούτως ώστε να δουν αν θα μπορέσουμε να πετύχουμε αυτό το στόχο. Αν πάντως εξετάσουμε τα οικονομικά προβλήματα τα οποία σοβούν, θα πιστούμε ότι τα ίδια θα έχει να αντιμετωπίσει και η επομένη Προεδρία. Η Δανέσικη Προεδρία επίσης θα ασχοληθεί και με τους προπολογισμού με τη μεσονική πολιτική της περίοδου 2010-2020. Θα χρειαστούμε περισσότερους πόρους για την ανάπτυξη των νέων κρατών μέλων. για και ανάπτυξη θέλει η Δανειακή Προεδρία. Ταυτόχρονα όμως θα πρέπει να προσέξει την δέσμη μέτρων για την αλλαγή του κλίματος. Διακόπτη Πρόεδρος. Ε, κυρία Πρωθυπουργέ, εύχομαι να έχει επιτυχία η Προεδρία σα. Βέβαια η εξάμηνη εκπεριτροπή Προεδρία έχει μείζωνα συμβολισμό της δημοκρατικής λειτουργίας της ευρωπαϊκής ένωσης. δεν αφήνει όμως περιθώρια ουσιαστικής επίδρασης στα πράγματα. η χρονική περίοδος της εξάμηνης δανεικής προεδρίας συμπίπτει με χρόνο αποφασιστικό για το μέλλον της ευρώπης και των πολιτών της. είναι σαφές ότι τα θεσμικά όργανα της ένωσης έχουν υποκατασταθεί από ένα άτυπο διευθυντήριο το οποίο δεν έχει επιτύχει. ελπίζουμε ότι ο νέος πρόεδρος κ. σουλτς τον οποίο επιλέξαμε χθε θα προσπαθήσει να ανατρέψει αυτή την κατάσταση. η ελλάδα κυρία ε, πρωθυπουργέ είναι απόδειξη της αποτυχίας της οικονομικής πολιτικής της ευρώπης και συνακολουθείται από την ιταλία και όλες τις άλλες χώρες του νότου. η λιτότητα έχει αποτύχει η ανεργία έχει απογειωθεί τα ελλείμματα αυξήθηκαν η ύφεση γιγαντώθηκε και περιπέσαμε τελικά σε κατάσταση ε, ιστορικής παγίδας. Πράξτε να βελτιωθεί η κατάσταση. Ευχαριστώ και τώρα το λόγο έχει η συνάδελφος Άουκεν. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Να ευχαριστήσω και τον, ε, την Πρωθυπουργό η οποία έκανε μια πολύ καλή ομιλία, μας κάνει υπερήφανους. Μία ερώτηση θέλω να θέσω στην Πρωθυπουργό για το άρθρο 41 του χάρτη για την καλή διακυβέρνηση. Πρόκειται για κάτι το οποίο απασχολεί και τους πολίτες αλλά και τα θεσμικά όργανα. Δεν λαμβάνουμε τέτοιες ε, νομοθεσίες για την ε, χρηστή διακυβέρνηση. Ίσως θα χρειαστεί από πλευράς της ε, να δοθεί μια μικρή πίεση. το άρθρο 41 για την ε, χρηστή διακυβέρνηση θα πρέπει να εισαχθεί. Θα σας ζητούσα λοιπόν να το πράξετε αυτό. Δεν είναι ίσως τόσο ενδιαφέρον το θέμα, αλλά είναι πολύ σημαντικό. Η κυρία Κονή. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Συγχαρητήρια. Η απασχόληση σε αυτή την κρίση που περνάμε κυρία Πρωθυπουργέ πρέπει να αποτελεί προτεραιότητα. 23 εκατομμύρια επιχειρήσεις έχουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση και αντίστοιχους ανέργους. Κάντε την εξίσωση. Πρέπει λοιπόν να συνεργαστούμε για να μπορέσουμε να δώσουμε στους πολίτες μας το κέφι να ξεκινήσουν ξανά να επιχειρούν Πρέπει να δει λοιπόν η Κομισιόν πώς θα προχωρήσει τις κοινωνικές επιχειρήσεις 100 δισεκατομμύρια ευρώ μπορεί να αντιπροσωπεύσει στην Ευρωπαϊκή Ένωση και 7,5% των ευρωπαϊκών εργατικών χεριών. Είναι μια φιλόδοξη πρόταση κυρία Μπαρόσο, εύστοχη πρόταση και θα ήθελα μαζί κυρία Πρωθυπουργέ να μπορέσουμε να εγκρίνουμε την οδηγεί αυτή κατά τη δική σας Προεδρία. Ευχαριστώ κυρία Κονή και το λόγο έχει ο συνάδελφος Ταχτάν. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ για το πρόγραμμά σας. Κατά το τελευταίο εξάμεινο ή το Κοινοβούλιο εκπώνησε μια έκθεση για την καταπολέμηση της στόχιας. Βλέπουμε το φαινόμενο όμως να οξύνεται εδώ στην Ευρώπη και αυτό λόγω των μέτρων λιτότητας που λαμβάνονται στα διάφορα κράτη-μέλη. Ενώ λέγεται σαφώς ότι τα μέτρα αυτά δεν θα έπρεπε να πλήξουν τον κοινωνικό ιστό και την απασχόληση. Ποιο τι θα κάνει η Προεδρία σας για να ενθαρρύνει τον κύριο Άντορ ούτως ώστε να συνεχίσει τις πολιτικές για τη μείωση της φτώχειας και των φτωχών στην Ευρώπη. Η έκθεση συστήνει να δοθεί μεγαλύτερη δημοσιονομική υποστήριξη στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα για την καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού και της φτώχειας. Πώς βλέπετε εσείς να υλοποιείτε αυτή η σύσταση μέσα στο πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο. τι συγκεκριμένα μέτρα, ας πούμε παράταση μετά το 2013 για την επιστημική βοήθεια υπέρ των φτωχών, αυτά τα προγράμματα διακυδεύονται σε επίπεδο ορισμένων χωρών. Ευχαριστώ κύριε συνάδελφε Νταρντάν και τώρα από την πλευρά της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για να απαντήσει ο Επίτροπος Μπαρόσο. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Τα ερωτήματα αυτά όλα απευθύνθηκαν στον Πρωθυπουργό, στην Προεδρεύω να του Συμβουλίου. Δεν πρόκειται λοιπόν να τις αφαιρέσω αυτό το πλεονέκτημα να απαντήσω στις ερωτήσεις. Θα ήθελα όμως να επαναλάβω την ανάγκη να επικεντρωθούμε για να συμπληρώσουμε τις σημαντικές μας προσπάθειες σε ό,τι αφορά τη δημοσιονομική ολοκλήρωση με μέτρα ανάπτυξης. Και πιστεύω ότι η Δανική Προεδρία θα είναι ένα πάρα πολύ αποτελεσματικός εταίρος σε αυτό το πλαίσιο για ε, την εξέβρεση πραγματικών ε, λύσεων. Νομίζω ότι, κυρία Πρωθυπουργέ, υπάρχει ευρία υποστήριξη από πλευρά του Κοινοβουλίου για το πρόγραμμά σα. Μπορείτε να υπολογίζετε στο Κοινοβούλιο, μπορείτε να υπολογίζετε ασφαλώ και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, προκειμένου να μην ε, καταστεί αυτό το εξάμεινο, εξάμεινο καθυστερήσεων, αλλά ε, εξάμεινο συγκεκριμένων ε, μέτρων. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε Μπαρόσο. Και τώρα η κυρία of Σμιτ. Uh, κύριε Πρόεδρε, κύριε Πρόεδρε της Επιτροπής, εξωτήμοι βουλευτές, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τις παρατηρήσεις σας. Για μένα ήταν ε, πραγματικά αιτία ικανοποίηση το να συμμετέχω σε μια τέτοια συζήτηση όπως η σημερινή. Αυτό το οποίο κρατώ από τη σημερινή συζήτησή μας είναι ε, το ότι ναι, όντως δεν μπορούμε όλοι να συμφωνήσουμε, όμως ε, η εντύπωσή μου είναι ότι επιβεβαιώνεται με τρόπο πανηγυρικό ότι πρόκειται να στηρίξετε το πρόγραμμα της Δανικής Προεδρίας και σας ευχαριστούμε γι' αυτό. Θα κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας, ούτως ώστε να σταθούμε στο ύψος των ε, περιστάσεων και να εμφανούμε εντάξει της εμπιστοσύνη σας, πιέζει ο χρόνος. Βεβαίω, ε, αλλά θα πρέπει να σταθώ σε κάποια από τα σημεία τα οποία θίξατε. Κύριος Μπάρος και ο κύριος ε, Ντάου ε, είπατε για το θέμα του IFF. Βεβαίως και πάρα πολύ σοβαρά θα ασχοληθούμε και με αυτό το θέμα κατά την Προεδρία. Για να μπορέσουμε το πολιτές μεσονομικό πλαίσιο να πλαισιωθεί όπως πρέπει και να εξυγχρονίσουμε τις δημοσιονομικές προοπτικές. Να εμπιστατεύσουμε τους κοινούς πόρους για δημιουργία θέσεων εργασία και ανάπτυξης. Επίσης, να σας πω κάτι σε σχέση με αυτό το οποίο είναι ο και άλλες για τον ε, φόρο των χρηματοπιστωτικών συναλλαγών. Θα αυτό θα ήθελα να σας το πω, ούτω να διασκεδαστούν κάθε φόβη και αμφιβολίες. Η Δανέζικη Προεδρία πρόκειται να διεκπεριώσει ε, το θέμα αυτό ε, όσο πιο ξεκάθαρα όσο πιο τίμια μπορεί. Θα πρέπει να δούμε τι θα γίνει με το σχετικό κανονισμό, ούτω ώστε να μπορέσουμε να ενισχύσουμε το ρόλο τη κοινότητα και την Προεδρία μα. Πάρα πολλοί επίση στάθηκαν στο πρόβλημα τη Προεδρία Φερχόφστατ Χάρμς, αλλά και ο κύριο Μωράε ε, το σχολίασε. Όπω όλοι γνωρίζετε, τώρα, ε, σήμερα κιόλα, το θέμα θα συζητηθεί στην Ολομέλεια, αλλά πάντως μπορώ να σας πω με λίγα λόγια ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διαδραματίζει πάρα πολύ σημαντικό ρόλο. Είναι ο φύλακα των συνθήκων και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα αρχίσει τη διαδικασία επί παραδιάση της ε, ε, συνθήκης επί τη βάση τριών ε, λόγων, τριών άρθρων. Και εμείς θα στηρίξουμε την πρωτοβουλία της ε, Ευρωπαϊκής Επιτροπής γιατί ακριβώς πρόκειται για τους κανόνες που έχουμε στα χέρια μας και την κοινωνική μέθοδο. Επομένως δεν μπορούμε να παρασταθούμε στο πλευρό της Επιτροπής για το θέμα τούτο. Και όλοι πρέπει να συμμορφωθούμε με το κείμενο δίκαιο. Διότι έτσι λειτουργεί η Ευρωπαϊκή Ένωση. Πάρα πολύ. επίσης ανέφεραν την κρίση την ε, υποβάθμιση από του οίκου αξιολόγηση πολλών χωρών. Τι απαντήσει πρέπει να δοθούν σε πάρα πολλά ερωτήματα για αυτή την κρίση. Όμω, πριν απ' όλα, πριν θεωρήσετε ότι πρόκειται για κρίση που σοβεί στην Ευρώπη. Σα υπενθυμίζω ότι ο λόγο τον οποίο φτάσαμε σε αυτή την κρίση εδώ στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ο λόγο είναι το ότι τα κράτη-μέλη δεν φρόντισαν όπω θα έπρεπε τα δημοσιονομικά του. Γι' αυτό έχουμε το πρόβλημα. Άρα Εκεί να επικεντρώσουμε προσοχή μα και να βρούμε φυσικά ευρωπαϊκέ πανευρωπαϊκές λύσεις αλλά να μην ξεχνούμε τι αιτίε τη κρίση. Τα κράτη-μέλη τα οποία δεν ετήρησαν κάποιου κανόνε. Και τώρα όσον αφορά την υποβάθμιση των οικονομικών κρατών μελών, αυτό είναι κάτι το οποίο το ανέφερε και ο κύριος ε, Φερχόφστατ, που μνημόνευσε και την ε, Standard and Poor's πάρα πολύ συγκεκριμένα αναφέρθηκαν στην ε, έλλειψη προοπτικών ανάπτυξης και προέβησαν στην υποβάθμιση κάποιων χωρών. Δεν το είπε ε, κάποιος αριστερός, κάποιος σοσιαλδημοκράτης. Το είπε η Standard Poor's. Ότι δηλαδή η λιτότητα θα πρέπει να πηγαίνει χέρι-χέρι με ανεπτυξιακές πρωτοβουλίες. Οπότε και ερχόμαστε στη συζήτηση σε σχέση με απασχόληση και ανάπτυξη, κάτι το οποίο το ανέφεραν πάρα πολλοί, Σφόμποντα, Χάρμς, Σόργαρντ, Τόρενσον, Μπένσον και άλλοι από τους αγορητές. Οπότε, θα πρέπει ξεκάθαρα να σας πω ότι η οικονομία της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα πρέπει να ενδυναμωθούν η Προεδρία, η Δανία. Ακριβώς τέτοια πολιτική θέλει να ασκήσει. Όμως δεν αρκεί, δεν αρκεί το νοικοκύρεμα των δημοσιονομικών. Θα πρέπει να υπάρξει και μια όθηση των οικονομιών προς ανάπτυξη και απασχόληση. Αυτό περιμένουμε από εμάς όλοι και κυρίως οι νέοι να δημιουργήσουμε απασχόληση στην Ευρωπαϊκή. Συμφωνία με όσου λόγο και είπαν ότι ίσως θα πρέπει να θυμηθούμε ε, μία από τη μεγαλύτερη μας ε, επιτυχία ίσως η πιο μεγάλη που ήταν η ενιαία αγορά η οποία δημιούργησε και απασχόληση και ανάπτυξη και να συνεχίσουμε να ολοκληρώσουμε τη διαδρομή της ε, ενιαίας αγοράς ο πρώτος του Συμβουλίου και εγώ είπαμε ότι δεν θα πρέπει να διστάσουμε μπροστά σε μια τέτοια κατεύθυνση και στις 30 Ιανουαρίου που θα έχουμε τη συνάντηση κορυφή, θα το συζητήσουμε με έμφαση το θέμα. Οπότε θα συζητήσουμε όχι μόνο τα, του νοικοκυρέματο των, των δημοσιονομικών, θα συζητήσουμε, θα συζητήσουμε και τα τη ανάπτυξη και τα τη απασχόληση. Πάρα πολύ. Από σα επίση αναφέρετε την ε, οδηγία για την ενέργεια, την, ε, την, την ε, αποτελεσματική της χρήση. Κύριε Τούρμες, σας ευχαριστώ που το είπατε και σας τονίζω ότι αν θέλουμε να έχουμε αυτά αποτελέσματα για τα θέματα του περιβάλλοντος θα πρέπει να δουλέψουμε κατεπηγόντως. Έχουμε την ευκαιρία. Ε, έχουμε το Κοινοβούλιο που συμφωνεί, έχουμε την Προεδρία που επίση θέλει να κάνει κάτι τέτοιο. Επομένω, α πάμε προ εκείνη την κατεύθυνση για το επόμενο εξάμεινο. Και αυτό θα το πετύχουμε μόνο εάν συνεργαστούμε. Επίση, πολύ εξημώνα αναφέρατε την ενότητα, την κοινοτική μέθοδο. Και σας ξεκαθαρίζω ότι αυτό το οποίο κάνει η Ευρώπη να ξεχωρίζει είναι το ότι έχουμε δεσμευτεί να είμεθα αλληλέγγυοι, να είμεθα ενωμένοι, αλλά επίσης το ότι απαρέγκλητα θέλουμε να ισχύει η κοινοτική μέθοδος. Όσοι ακούν αυτή τη συζήτηση θα μπορούσαν να απορρίσουν τι πάει να πει η κοινοτική μέθοδος. Όχι, πρέπει να συνεχίζουμε να την πρεσβεύουμε και να την προωθούμε την ε, γενική μέθοδο, διότι Ευρώπη σημαίνει ότι δεν πριτανεύει το δίκαιο του ισχυρού. Στην Ευρώπη έχουμε κράτος δικαίου και πριτανεύει η δημοκρατία και αυτό ακριβώς και θα πρέπει να συνεχίσουμε να προστατεύουμε. Και αξίζει και όχι μόνο για χάρη των ε, μικρότερων αλλά για χάρη όλων η ενότητα και η κοινωνική μέθοδος θα πρέπει να είναι ο υπέρτατος στόχος και να διέπει όλες μας τις προσπάθειες. Οπότε σας παρακαλώ, ε, πρώην συνάδελφοι, φίλοι, ε, μέλη του Κοινοβουλίου, όλα αυτά ας τα υλοποιήσουμε, ας συνεργαστούμε και ας ε, πετύχουμε κάποια απτά αποτελέσματα για χάρη των Ευρωπαίων. Εγώ είμαι πεπισμένο ότι μπορούμε να τα καταφέρουμε. Και αν τα καταφέρουμε θα ανοίξουμε το δρόμο ούτω ώστε να υπάρχει κάποια διέξοδο και να έχουμε ένα μέλλον με περισσότερη ευημερία. Σα ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε του Συμβουλίου. Σα ευχαριστώ, κύριοι συνάδελφοι, για την πειθαρχημένη σα ε, παρέμβαση. Θα σα παρακαλέσω να κάτσετε τώρα, προκειμένου να συνεχίσουμε με την ημερήσια διάταξη.